ορίσαμε την πολιτική μας ε, προσέγγιση στο θέμα της σήμασης στον τομέα της κλωστοϊφαντουργίας και δεν θέλουμε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης, θα γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια καταρχήν. Συμφωνία η Επίτροπη στην ε, πλήρη σύνθεσή της. Μάντερς θα το διαβιβάσει στο Συμβούλιο. και θα γίνει ψηφοφορία πρώτης ανάγνωσης το Μάιο 1 ή 2. Επίσης, η προφορική μας ερώτηση ως προς ε, τις αλλαγές από πλευράς ε, καταναλωτή, καταναλωτών, η πρότασή μας έγινε αποδεκτή και θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο τμήμα της μήνυ ολομέλειας των Βρυξελών. Αυτά ήταν τα σημεία. Η κυρία Ρούλε κάτι ήθελε να μας πει για το χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού. Της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλές φορές ε, είπα να προσέξουμε ότι αυτή τη χρονιά δεν είχαμε πολύ χρόνο για να προετοιμάσουμε τον προπολογισμό όπως κατά το, παρελθόν. Ε, οι προθεσμίες από την Επιτροπή Προπολογισμών είχαν οριστεί για 12 Μαΐου και ε, θα μπορούσε κανείς να συνεργαστεί με τους σκιώδεις ε, εισηγητές των διαφόρων ομάδων. 12 ε, Μαΐου θα παρουσιαστούν οι τροπολογίες στην Επιτροπή μας. Θα σας προτείνω λοιπόν να συναντηθούν οι σκιώδεις ε, εισηγητές 11 Μαΐου για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Και να πω και κάτι άλλο. Μιλούμε για δύο-τρία πιλωτικά προγράμματα. Μιλούμε για το Solvit, για την ενιαία αγορά και το Forum. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Και πρέπει να μπορούμε να υποβάλουμε και τις κατάλληλες ε, τροπολογίες έτσι ώστε να μην υπονομευθεί η θέση μας. Ευχαριστώ. Για τον προπολογισμό, κυρία Στάτλερ, ωραία, να δούμε τα, του προπολογισμού πρώτα και μετά τη δική σας ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, όπως προτείνει η κυρία Ρούλερ, θα προχωρήσουμε. Οι ομάδες και οι σκιώδες σας να αντιθούν για να συνεχιστεί η διαδικασία. Η κυρία Στάτλερ ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή ΕΚΟΝ τώρα ψηφίζουν για την ε, οδηγία για, τις, ε, για τα μηχανοκίνητα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε και εμείς ποιο θα είναι το, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι το ψήφισμα για να κοινοποιηθούν οι απόψεις του Κοινοβουλίου ήταν η δική μας ιδέα ούτως ή άλλως. Οπότε χαίρομαι που τα κατάφερε η ΕΚΟΝ και υιοθέτησε την απόψή μας, ε, παρόλο που είναι μόλις ένας μήνας μέχρι να τεθεί σε ισχύ το ψήφισμα. Από τον προηγούμενο Οκτώβρη την έχουμε κάνει με την πρόταση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα υπάρξει βέβαια και άλλη δυνατότητα, γιατί ούτω ή άλλω πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το ψήφισμα από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Οι συνάδελφοι λοιπόν που, ενδιαφέρουν, που του ενδιαφέρουν τα θέματα καταναλωτών μπορούν να πούν την απόψη του. Ευχαριστούμε την κυρία Στατλέρ που μα το θύμισε. Προχωρούμε. Πάμε στην έκθεση του κυρίου Γκρέγκ για την ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Κάναμε εντατικές συζητήσεις και ενδελεχείς με τον καθηγητή Μάριο Μόντι, ο οποίος εργάζεται παράλληλα και σε άλλη μία γνωμοδότηση. Ο κύριος Γκρέκ έχει λάβει 236 ε, τροπολογίες. Η χρονική στιγμή της ε, γνωμοδότησης αυτής φαίνεται ότι είναι η πιο σωστή, γιατί η έκθεση του κυρίου Μόντι θα, υπο, θα δημοσιευθεί κάπου κοντά και με τη δική μας έκθεση. Οπότε, να δώσω στον κύριο Γκρέκ την, ε, το λόγο για να μιλήσει για τις ε, τροπολογίες και μετά οι σκιώδεις. Δεν ξέρω τώρα ποιος εκπροσωπεί το ΕΛΚ. Ο κύριος Κάρας ψηφίζει στην ΕΚΟΝ, οπότε ο κύριος Ρόσφολ είναι εδώ. Ο κύριος... Ε, η κυρία είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Ο κύριος Ντιγιόν επίσης είναι εδώ. Ωραία. Οπότε, πρώτα στους κοιόδες, ο λόγος. Καλωσορίζω και την κυρία Μπρόμπτο που ήρθε. Κύριε Γκρέκ, πριν ξεκινήσετε, να πω ότι γίνεται μετάδοση στο ίντερνετ της συνεδρίασής μας, οπότε παρακαλώ χρησιμοποιείτε το αριστερό μικρόφωνο για να σας παίρνει πιο καλά η κάμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. 236 τροπολογίες έλαβα. Από όλους. Προσπαθώ να δω πώς θα τα συμβιβάσω όλα. Γιατί πραγματικά είναι πολλά τα αιτήματα των ομάδων. Παρ' όλα αυτά, να πω εξ αρχής ότι δεν θα μπορούσα να επιτρέψω να γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο η έκθεσή μου. Έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένο για παράδειγμα, ένα θέμα που είχα ήταν ο τίτλος «Μια ενιαία αγορά για τους καταναλωτές και τους πολίτες». Δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι αποκλείω τις τέσσερις ελευθερίες ή τα άλλα, τις άλλες οικονομικές πτυχές της ενιαίας αγοράς. Αλλά αν έπρεπε να τα συμπεριλάβω όλα, προφανώς δεν θα τέλειωνε ποτέ η έκθεσή μου. Για παράδειγμα, δεν αναφέρω τι επιχειρήσει, γιατί αν δείτε την έκθεση, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω τι επιχειρήσει. Μίλησα για τι μικρομεσαίε, έγραψα λίγα πράγματα για τι μικρομεσαίε, αλλά αν έπρεπε να μιλήσω για τι επιχειρήσει, δεν θα συνδεόταν αυτό με τίποτα πώ αναφέρεται στην έκθεση. Θα ήταν ξεκρέμαστο. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οι επιχειρήσεις στην έκθεση, αλλά δεν γινόταν να γίνει σε αυτή την έκθεση. Γιατί αλλιώ θα αντίκειτο όλο αυτό στο βασικό στόχο τη έκθεσή μου. Τις περισσότερες από τις τροπολογίες τις έχω συζητήσει με τους σκιώδεις. Έχουμε πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και δουλεύουμε αρκετά καλά. Αρκετά λογικά προχωρούμε και από χρονικής πλευράς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να συζητήσω και με άλλους σκιώδεις. Να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία για να ικανοποιηθούν όλες οι ιδέες. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Απ' την άλλη πρέπει να στείλουμε και ένα σαφές ε, πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα αναζωογονηθεί η ενιαία αγορά και δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε μια έκθεση συγκεκριμένη και όχι μια αναποτελεσματική έκθεση. Οπότε θα συνεχίσω να είμαι στη διάθεσή σας για τα σχόλιά σας ε, κύριε Σκιώδης. Πάντα χαίρομαι να ακούω τα σχόλια των συναδέλφων και περιμένω τα σχόλιά σας σήμερα, αλλά πρέπει να τονίσω ότι η έκθεση πρέπει να είναι στοχοθετημένη, πρέπει να είναι συγκεκριμένη, δεν μπορούμε να βάλουμε νερό με απόψεις, ε, ακόμη και από τη δική μου την ομάδα, έπρεπε να απορρίψω κάποιες ε, αιτήσει ε, για προσθήκε. Οπότε ζητώ την κατανόησή σας, γιατί ήταν δύσκολη η δουλειά αυτή. Θα κλείσω εδώ τα σχόλιά μου και βεβαίως μετά θα ακούσω με ευχαρίστηση τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λουί. Uh, um, λοιπόν, όντω πρέπει να είναι πολύ στοχοθετημένη η έκθεση γιατί έχουμε και κάποιε συστάσει κλειδιά. Πρέπει να είναι σημαντική ε, σημαντικές οι συνέπειες που θα προκύψουν από την ε, έκθεσή μας. Πρέπει να δώσουμε σαφώς το στίγμα μας και προς το Συμβούλιο και προς την Κομισιόν. Ελπίζω λοιπόν ότι όλες οι ομάδες θα συνεργαστούν προς αυτό το σκοπό. Και έχω και την αίσθηση ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Και με χαροποιεί αυτό βεβαίω. Να είμαστε προσεκτικοί, να μην συμπεριλαμβάνουμε πράγματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο, στην δική μας την εντολή εδώ, της Επιτροπής μας. Είναι ε, έκθεση της Επιτροπής αυτή. Δεν είναι ψήφισμα για την Ευρώπη του 2020, που υπάρχει ούτως ή άλλως, οπότε καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στις βασικές συστάσεις. Βέβαια, οι πολιτικέ ομάδε θα το αποφασίσουν αυτό, αλλά η δική μου πρόταση αυτή είναι. Ελπίζω να μπορείτε να τη δεχτείτε. Ο κύριος Κάρας δεν έχει έρθει, οπότε ας προχωρήσουμε στον κύριο Ρόσφορ, την κυρία Ρουλέ, μετά θα μιλήσω εγώ για την ομάδα μου, ο κύριος Διόν, και αν έχει έρθει και ο κύριος Κάρας θα τον ακούσουμε. Θα δώσουμε το λόγο και στην κυρία Γκέπχαρτ ο κύριος Ροσφόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κρέσ για το έργο του που έκανε για μας 236 ε, τροπολογίες είναι για όλους εμάς. Ε, εμείς δηλαδή τις προκαλέσουμε και πραγματικά δουλεύετε σε περιορισμένο χρόνο και χρονοδιάγραμμα. Όταν έχουμε τόσες τροπολογίες σε ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει να καταλάβει κανείς γιατί για μένα είναι το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα σε ορισμένους συναδέλφους να υπάρξει μια ισορροπία σε τέτοιο κείμενο. Σε σχέση με το διάλογο που είχατε θα έπρεπε να είναι σαφές ότι αυτός ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει ένα σωστό παράδειγμα της κρίσης που έχουμε στην εσωτερική αγορά. Ότι έχει κουραστεί η εσωτερική αγορά. Από τη στιγμή που έχετε ένα κείμενο που δίνει έμφαση στον καταναλωτή και τον πολίτη, η, η επικυρότητα, η συγκυρία που βλέπουμε οικονομική σήμερα, Αυτό είναι και ο αρχικός σας τίτλος. Δηλαδή, από τη μια μιλάτε για την εσωτερική αγορά για να καταλήξετε στον πολίτη. Αυτά μας κάνουν να καταλάβουμε και να δώσουμε την εξήγηση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά δηλαδή ότι υπάρχει η επιθυμία ε, ειλικρινής από πολλούς ε, ευρωβουλευτές να θίξουν κάποια θέματα και να δούνε τους στόχους που έχετε κι εσείς αναφέρει. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα λοιπόν που αφορά εμένα και την ομάδα μου. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες όπου ξαναθίγουμε το θέμα της αναγκαιότητας να αναφερθούν πολύ, να δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διότι η φύση της εσωτερικής αγοράς είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά η οποία είναι ανισόρροπη. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα που πρέπει να γίνει για να δει κανεί ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα σε συμφέροντα του πολίτη, καταναλωτή και αυτά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ, σαν θέση, είχα το εξή. Να σα προτείνω τροπολογίε που θίγουν αυτό το θέμα, αυτή την πτυχή και κυρίως στα κεφάλαια που αφορούν τον πολίτη και καταναλωτή. Εκεί ας πούμε δεν θα αναφέρουμε τροπολογίες που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή να είμαστε σαφείς τους στο στόχο μας. Δηλαδή ε, να μην επανερχόμαστε σε κεφάλαια με διαφορετικής φύσης τροπολογίες. Έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο φυσικά είναι πολύ αυστηρό, το καταλαβαίνουν όλοι εδώ και όλοι πραγματικά θέλουμε να είμαστε πιστοί στις προθεσμίες μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και στις προσδοκίες όλων. Να πω ότι, παρόλα αυτά, ότι έχουμε κάποιες δυσκολίες. Από τη στιγμή που μιλάμε και αύριο θα έχουμε ψηφοφορία, εγώ δεν έχω τη μετάφραση αυτών των 236 τροπολιών στη γλώσσα μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τους άλλους συναδέλφους δεν θα ήθελα να πω, εντάξει όλες οι γλώσσες έχουν σημασία, αλλά, αλλά να μην έχω τώρα εγώ τη μετάφραση στη γλώσσα μου, ε, πραγματικά να μην κάνω τώρα μια απειλή, αλλά δεν είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε για ψηφοφορία. Καταλαβαίνουμε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ δύσκολο. Για παράδειγμα, όταν έχουμε τόσες απολογίες, 236, δεν ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοι, πρέπει κανείς να τις δει κανείς αυστηρά στο μικροσκόπιο την κάθε μία. Υπάρχουν τροπολογίες όπου ζητώ να διαγραφούν κάποιες φράσεις. Όχι ότι διαφωνώ με τη βασική ιδέα της φράσεως, αλλά διότι βλέπω ότι ξαναεπανέρχεται αυτή η φράση λίγο αργότερα κάπου αλλού. Θα πρέπει λοιπόν να, πρέπει, να υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό τροπολογιών και να μπορεί κανείς να ελέγχει, να καταλαβαίνει πώς ακριβώς έχει το κείμενο. Όταν έχει λοιπόν τόσε πολλέ τροπολογίε, δεν έχει το χρόνο κανεί να μπορέσει να ελέγξει, φέρει πίν, αν ε, η α ή β φράση σε μια τροπολογία επανέρχεται κάπου αργότερα. Και να κλείσω λέγοντας ότι συμφωνώ μαζί σας και οι δύο ότι σε ένα τέτοιο θέμα θα πρέπει πάντοτε να πετυχαίνουμε μια συνένεση. Εγώ από τη δική μου μεριά θα κάνω τα πάντα και νομίζω πάρα πολλοί εδώ μέσα θα σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Τόσο στι συμβαστικέ τροπολογίε πάνω στις οποίες δουλεύετε ε, σήμερα και θα συνεχίσουμε φυσικά και αύριο. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριο Ρόσφορ. Δεν είναι διαθέσιμες οι τροπολογίες, το γνωρίζουμε και η Γραμματεία προσπαθεί να τις προωθήσει το ταχύτερο δυνατόν. Ε, χαίρομαι όμως ότι συνεργάζεστε υπό τόσο δύσκολες συνθήκες και σε ένα τόσο αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Κατανοούμε τη σημασία της έκθεσης αυτής. Θα πρέπει να συζητηθεί μαζί με την πρόταση της Επιτροπής και την έκθεση του κυρίου Μόντε. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μπαρνιέ που θα έρθει στην ακρόασή μας σήμερα το απόγευμα ως προς το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με την έκθεση Μόντι. Και θα το συζητήσω με τον εισηγητή. Θα πρέπει όμως να ψηφίσουμε αύριο έτσι ώστε να έχουμε μία δήλωση ενώπιν Σολομέλιας. Ρούλε. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Ένα σημείο μόνο θα ήθελα να τονίσω. Οι 236 τροπολογίες δεν ε, μιλούν μόνο για την κρίση της εσωτερικής αγοράς, μιλούν και για, την, ε, για τα ιδιωτικά συμφέροντα που υπάρχουν στην ε, εσωτερική αγορά. Οπότε θα ήθελα να σας πω, να πω μάλλον στον εισηγητή, ότι έχω μεγάλο ενδιαφέρον να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι δεν έχει νόημα να βάλουμε νερό στο κρασί μας μέσω διαφόρων φέσεων που προκύπτουν από κάποιες τροπολογίες. Γιατί αλλιώ δεν θα επηρεάζουμε τα πράγματα. Ε, θα υπάρχει και η έκθεση μόνη για την εξέλιξη τη εσωτερική αγορά. Οπότε η, πραγματικά μεγάλο σεβασμό έχω για την δουλειά που κάνατε και όντω συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να δώσουμε ένα συγκεκριμένο α, μήνυμα. Ε, κάντε λοιπόν ό,τι μπορείτε να καταλήξουμε συμβασμού για να μην χρειαστεί να βάλουμε νερό στο κρασί μα. Uh, well, if, um, I would perhaps contribute... Ω κοιόδη, θα ήθελα να πω και εγώ ορισμένα πράγματα για την ομάδα μου. Καταρχήν συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι με τον κύριο Κρέχ για το ότι θα πρέπει να προβάλλουμε μια δυναμική θέση. Με ενθαρρύνεται ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την έκθεση, γιατί πολλές φορές ε, θεωρούν ε, οι ενδιαφερόμενοι ότι οι εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας δεν είναι ύψης της σημασίας και ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει το μεγάλο σας ενδιαφέρον. Συμφωνώ με τον κύριο Ροσφόρ ότι ίσως υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή μας δεν θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ε, βρίσκεται πρώτων πυλών. Υπάρχουν πολλά ζητήματα για προέκτασή της προς τους πολίτες, και τους καταναλωτές. Η έκθεση του Λουί προβάλλει πολλές προτάσεις και συνεισφέρει εμπολής προς αυτή την κατεύθυνση η έκθεση αυτή. Με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στοιχεία για τις ε, ΜΜΕ. Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Λουί, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλοί πολίτες είναι μικροεπιχειρηματίες και αυτό προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλουμε να αρχίζουν ε, τις εργασίες τους νέες μικροεπιχειρήσεις και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στην οδηγία περί Είναι μια οδηγία η οποία ε, θέλει να προβάλλει πληροφορίες για τις ΜΜΕ έτσι ώστε να ε, δράτουν ευκαιρίες εκεί όπου μπορούν. Και ένα ιδιαίτερο σημείο αφορά ένα σημείο, ένα θέμα δράσης που ο Λουί Κρέκ έθεσε υπόψη για ένα νομοθετικό πακέτο. Νομίζω ότι πρέπει να το θεωρήσουμε ευρύτερα με βάση την πράξη περί ΜΜΕ, Small Business Act, η οποία θα συγκεράσει τα νομοθετικά και μη στοιχεία της έκθεσης του Λουί Κρέκ σε μία έκθεση ίδιας πρωτοπουλίας. Αυτή είναι μία από τις βασικές ιδέες που διέπουν αυτή την έκθεση και χαίρομαι διότι ο Λουί σε μία τροπολογία συμβασμού δίνει νέες διαστάσεις στο νομοθετικό σκέλος. Εάν μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία προβάλλοντας την Small Business Act με βάση αυτές τις πρωτοβουλίες και περιλαμβάνοντας ε, συγκεκριμένες δράσεις προς τα κράτη-μέλη, διότι πολλές φορές οι πολίτες δεν, δεν θεωρούν ότι αυτές οι πράξεις είναι προσπελάσιμες. Αν λοιπόν δώσουμε ένα, μια πολιτική διάσταση στο θέμα, θα έχουμε συνεισφέρει ουσιαστικά, έτσι ώστε το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια. Ενώ ένα νομοθετικό ε, πακέτο δεν θα είχε την ε, ίδια, τις ίδιες επιπτώσεις και τον ίδιο αντίκτυπο. Ελπίζω λοιπόν ότι ο Λουί θα εμψυχώσει αυτή την ιδέα στα πλαίσια του Small Business Act και θα συνεργαστώ με όλες τις πολιτικές ομάδες για να φτάσουμε σε ένα συνενετικό πακέτο που είναι κρίσιμο έτσι ώστε η έκθεση αυτή να έχει τον ε, πρέποντα αντίκτυπο. Ο κύριος Ντιγιόν έχει το λόγο. Uh, θα ήθελα να καταστήσω σαφές κάτι. Όταν είπα businesses, δεν μιλούσαμε για τις ΜΜΕ. Δηλαδή, δέχτηκα κάθε τροπολογία που σχετίζεται με τις ΜΜΕ. Όταν μιλούσα για επιχειρήσεις, δεν μιλούσα μόνο για τις μεγάλες. Δηλαδή, ε, δεν μπορούσα να εστιάσω την προσοχή σε όλες τις πτυχές της ενίας αγοράς. Όταν μιλάμε όμως για τις ΜΜΕ, μπορώ να δεχτώ, δέχτηκα τις περισσότερες τροπολογίες. Δεν υπάρχει καμία ένταση σε αυτό το θέμα. που είναι υπέρ των ΜΜΕ, όπως γνωρίζω. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς, όπως λέτε, λέτε. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω όλες τις ε, τροπολογίες που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Λούι Γκρέχ γιατί είναι πολύ σημαντική έκθεση και τον συγχαίρω διότι μπορεί και συμβάλλει σε μια έκθεση συνένεσης και όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι ιδέες του Λουί Γκρέχ ε, σε αυτή τη σημαντική έκθεση του πέμπτου πυλώνα ε, και ξέρουμε ότι είναι ένας πυλώνας τον οποίο έχουμε παραμελήσει τον τελευταίο καιρό. Σε μερικές τροπολογίες εμείς δίνουμε μια έμφαση στο πρόβλημα του στο ψηφιακό χάσμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θέλουμε να θίξουμε διότι οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ ε, αυτή την πτυχή. Ε, λένε ότι υπάρχει μεγάλο κόστος στη χρήση αυτού του μέτρου και θα πρέπει να το δούμε αυτό το πρόβλημα στην έκθεση που έχουμε. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία Υπό αυτή την πτυχή και θα το βρείτε μέσα στο κείμενο. Ένα δεύτερο στοιχείο στο οποίο εφιστώ την προσοχή είναι ότι στις βασικές τροπολογίες δεν είδαμε το θέμα ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε όσον αφορά τη, η λειτουργία του, της αγοράς έτσι όπως ακριβώ έχει κατάσταση. Έχει δοθεί, δοθεί πολύ προσοχή όσον αφορά στα ωφέλη τα βραχυπρόθεσμα, αυτό είναι σημαντικό, δεδομένο. Και είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε τα θέματα και μακροπρόθεσμα. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε σε αυτή την έκθεση. Και να δούμε πώς το μέλλον φέρει πίν να αποφεύγουμε την έμφαση όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμες ε, πτυχή και να δούμε φερπίν πώς ε, έχει να κάνει το θέμα με επιχειρήσει, οι οποίε έχουν, ε, βλέπουν τη βιωσιμότητα και πιο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Κατά τα άλλα, όπως έχετε καταλάβει, είμαι υπέρ αυτής τη εκθέσεω. είμαι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κάρα ήρθε. Θέλετε να λάβετε το λόγο αμέσως ή να δώσουμε το λόγο. Εντάξει, θα ακούσουμε αλλου δυο και μετά εσει Η κυρία Γκέπχαρτ, ο κυριο Σφάμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Λουί για την πραγματικά πολύ καλή δουλειά που έκανε. Ένα σημείο θα ήθελα που το έθιξε και ο κύριος Ροσφόρ για τις μεταφράσεις. Θα ήθελα να θυμίσω ότι πολλές ομάδες έχουν ζητήσει η, ε, να αναβάλλονται προς τα πίσω οι προθεσμίες για την υποβολή των τροπολογιών γιατί πολλές φορές δεν έχουμε τις ε, μεταφράσεις. Ζητήσαμε από τις ομάδες αν είναι σε θέση να εργαστούν μόνο με αγγλικά κείμενα. Οι ομάδες είπαν εντάξει και εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό, αλλά θα ήθελα απλώς να σας ευστήσω την προσοχή. Γιατί είχαμε ζητήσει την αναβολή της προθεσμίας για τις, υπο... για τις ε, τροπολογίες, γιατί πάντα προκύπτει το θέμα των μεταφράσεων. Για να είναι σαφή λοιπόν τα πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα αν είχα τα κείμενα στα γερμανικά, το καταλαβαίνετε. Αντί να κάθομαι τώρα να διαβάζω αγγλικά. Αλλά το κείμενο του κυρίου Γκρέχ είναι τόσο καλογραμμένο που ακόμη και στα αγγλικά μπορώ να το παρακολουθήσω. Το δεύτερο σημείο που επίσης θα ήθελα να σας θυμίσω είναι ότι ως συντονιστές όταν λάβαμε την απόφαση να ξεκινήσουμε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. ήταν σαφές ότι έπρεπε να θέσουμε ω στόχο ποια είναι η σημασία της εσωτερική αγοράς για τους πολίτες και τους καταναλωτές της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι έχουν ε, αποκλειστεί κάποια θέματα, σαφώ, αλλά είπαμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους πολίτες που πάντα μα ρωτάνε τελικά τι μας δίνει εμάς η Ευρώπη, τι μας δίνει η εσωτερική αγορά. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε εμείς ως Επιτροπή και γι' αυτό ο Λουί έπρεπε κάποιους τομεί που φυσικά για την εσωτερική αγορά είναι σχετική, να τους αποκλείσει. Ε, φορολογία, ε, νομοθεσία για τη φορολογία, ε, θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, Ακριβώς γιατί δεν ήταν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, με τις απαντήσεις που ζητούν οι πολίτες. Και φυσικά σας δίνω δίκιο κύριε Ροσφόρ όταν λέτε ναι αλλά η κατάσταση τώρα στην οποία βρισκόμαστε με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση, την οικονομική κρίση Φυσικά θα, ε, θα θέλαμε κι εμείς να δώσουμε μια απάντηση σε αυτά τα θέματα, αλλά ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι αν θέλουμε να δώσουμε απάντηση καταρχήν στο πρώτο ερώτημα που θέσαμε. Φυσικά είναι δύσκολο να συγκεραστούν όλες αυτές οι απόψεις, αλλά θα ζητούσα αυτό που είπαμε στην δική μας την Επιτροπή να μπορέσουμε τουλάχιστον να δώσουμε μια απάντηση στις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι, α, οι πολίτες. Κύριε Ροσφόρ, ευχαρίστω αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια δεύτερη έκθεση, παρόλο που έχουμε και την έκθεση της κυρίας Τούρν, ε, για την οικονομία. Εκεί είναι η οικονομία στην πρώτη γραμμή και φυσικά εκεί θα ασχοληθούμε κυρίω με τα θέματα τη οικονομία και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ερωτη... απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν την οικονομία. Νομίζω λοιπόν ότι με την έκθεση αυτή του κυρίου Γκρέχ έχουμε ε, επιτύχει πολλά και επίση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η οικονομική πολιτική και η πολιτική για του πολίτε δεν αντίκεινται η μία στην άλλη. Αλλά συνδυάζονται και μόνο μπορούν από κοινού να δώσουν μια καλή απάντηση στον λαό της Ευρώπης. Και ο Λουί νομίζω ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Και αν δω και τις τροπολογίες, νομίζω ότι έχει προχωρήσει με τον καταλληλότερο τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό που έχει κάνει και θα τον ενθάρρυνα να συνεχίσει στην άγουσα αυτή. Και να θέσω και ένα ερώτημα προς το ΕΛΚ. Χαίρομαι που είναι ο κύριο Κάρας και ο κύριο Σφάμπ εδώ και θα μιλήσουμε μετά από μένα. Γιατί έχω ένα ερώτημα που ε, πάντα εκρεμεί μεταξύ των δύο ομάδων μας. Εσωτερική αγορά και η πράξη για την εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να προσυπογράψουμε ε, για, ως, ως σημάδι, ως μήνυμα προς τους πολίτες της Ευρώπης ότι έχουμε υπόψη μας και προσπαθούμε να υπεραμενθούμε των συμφερόντων τους. Γιατί μιλούμε για τομείς όπου δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις εργασίας, όπου παράγονται οι περισσότερες υπηρεσίες και τα περισσότερα προϊόντα. Αλλά ήταν καλό νομίζω και το ΕΛΚ. Εντάξει, έτσι να, να έκανε λίγο πίσω ρε παιδί μου, να μας έδινε λίγο χέρι, να μας πει εντάξει συμφωνούμε κι εμείς να έχουμε την πράξη για, τις, για την εσωτερική αγορά. Δεν είναι αντίφαση στα θέματα της οικονομίας αυτό. Ε, είναι απλώς ένα μήνυμα πολιτικό προς τους πολίτες ε, ότι σκεφτόμαστε το δικό του συμφέρον όταν εδώ στην Ευρώπη χαράσουμε πολιτική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που ήμουν απόν στην αρχή. Έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να ψηφίσω. Θα πάρει και ο σκιώδης μας, ο κ. Κάρας, την, ε, το λόγο αμέσως. Ε, θα ήθελα εγώ καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Γκρέχη για τη δουλειά του. Πραγματικά με τις προσπάθειές του κατάφερε να καταλήξει σε μια πολύ ισόρροπη έκθεση. Σας είμαστε ευγνώμονες λοιπόν για τη δουλειά που κάνετε Έχουμε αποστείλει τα σχόλιά μας, έχουμε αποστείλει πολλές ε, τροπολογίες, προσπαθήσαμε να εμπλουτίσουμε την έκθεσή του και νομίζω ότι τώρα πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό αυτό που είπε η Εύλην, είναι οριζόντιο το έγγραφο αυτό. Γιατί κάνει και ο κύριος Μόντι μία έκθεση και ξέρουμε ότι και ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα ε, προγραμματίζει την επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς. Είναι καλό λοιπόν που ακούγονται όλε αυτέ οι απόψει. Πιστεύω ότι η έννοια ε, πράξη της, για την εσωτερική αγορά, ε, κατά το πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, ε, εντάξει, πολλή φιλολογία είχε μέσα και όχι πολλά πρακτικά πράγματα. Οπότε, σε κάποια σημεία θα θέλαμε ίσως το κείμενο να γίνει πιο σαφές. Φυσικά είναι σημαντικό το ότι στο κέντρο της πολιτικής μας είναι οι, πολιτικές, είναι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο συνάδελφος Κάρα ήδη έχει συζητήσει μαζί σα ε, κάποιε προτάσει μα. Νομίζω ότι και χθε το βράδυ βρήκατε και κάποιε συμβαστικέ ε, προτάσει για τι 22, 32, 33, 34 και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν τόσο δεκτικός στι απόψει μα. Ευχαριστώ κύριε Σουβάμπ. Ο κύριο Κάρα. Herr Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συγητά, και εγώ ζητώ συγγνώμη. Ήμουνα στην Επιτροπή ε, Οικονομικών και έπρεπε να είμαι στην ε, ψηφοφορία, γιατί ήμουνα εισηγητής για, την, ε, για τα οχήματα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γκρέχ που από την αρχή έδειξε ανοιχτό πνεύμα και ανοιχτή διάθεση. Οπότε ξέραμε από την αρχή με ποιε από τι συμβαστικέ λύσει τι οποίε καταλήξαμε θα, θα είχαμε ίσω πρόβλημα στην ομάδα μα. Εντάξει, υπήρξαν κάποιε διαφορετικέ απόψει, για κάποια σημεία βρέθηκαν, α... βρέθηκαν συμβιβασμοί ο κύριος, η κυρία Γκέφχαρτ, συγγνώμη, ε, συνεχάρει τον ε, εισηγητή γιατί έκανε μια ισόρροπη γνωμοδότηση και βρήκε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των οικονομικών πτυχών της εσωτερικής αγοράς και των πολιτών και των συμφερόντων τους. Ενώνονται λοιπόν αυτές οι δύο πτυχές. Φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν αντιφάσεις και αυτό ακριβώς είναι το θέμα. καταφέρνει η έκθεση να μην βάλει τους ε, ε, πολίτες σε ένα στρατόπεδο και τις επιχειρήσεις σε ένα άλλο και να πολεμούν οι μεν τους δε. Α, ε, τέτοιου είδους ε, προβλήματα δεν θέλουμε να έχουμε, γιατί δεν αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της εσωτερικής αγοράς. Γιατί είναι σαν να λέμε ότι θα δώσουμε μόνο ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά για τους πολίτες Μόνο όταν βάλουμε στο κέντρο του, στον πυρήνα της συζήτησης, τον πολίτη. Η εσωτερική αγορά είναι εσωτερική αγορά για τους πολίτες. Αλλά δεν αφορά μόνο τους πολίτες, απευθύνεται και σε άλλους. Εμέσως μεν, αλλά απευθύνεται και σε άλλους. Οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε σε, στο ποια ακριβώς ιστορική αγορά θέλουμε. Γιατί αλλιώς θα... δεν θα έχει λόγο ύπαρξη ο όρος εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει τις ελευθερίες, ενισχύει την απασχόληση. Και στους πολίτες τους οποίους απευθύνεται, τους θέτει στο, στο κέντρο. Δημιουργείται λοιπόν ένα μοντέλο και μέσω της στρατηγικής της Λισαβόνας με την ε, βιωσιμότητα, με την κοινωνική ε, οικονομία. Όλα αυτά είναι στόχοι ούτως ή άλλως που πρέπει να επιτύχει η ε, εσωτερική αγορά και που πρέπει να αναφέρονται σαφώς. Οπότε ας μην δημιουργούμε προβλήματα. Έχουμε την υποστήριξη της συνθήκης της Λισαβόνας, οπότε ας, έχουμε, ας, ε, ε, στόχο, ας θέσουμε ως στόχο την εντατικοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Είπαμε ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε μέσω της εσωτερικής αγοράς να εμπλουτίσουμε τις ελευθερίες. Έχουμε τέσσερις ελευθερίες οι οποίες όμως δεν αρκούν. Είναι η ουσία και ε, το γράμμα και το πνεύμα ουσιαστικά της εσωτερικής αγοράς, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και πέρα από αυτό. Δεν θέλω τώρα να δημιουργήσω εδώ πέρα προβλήματα, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η εσωτερική αγορά. Δεύτερον, θα πρέπει σαφώς να πούμε ότι πρέπει να έχουμε μία στρατηγική ε, ανακοίνωσης, κοινοποίησης των πράξεων προς τους πολίτες, ενημέρωσης, να μπορούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες, γιατί αυτό έχει προστιθέμενη αξία. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν πουλάνε ποτέ αυτό που κάνουν. Ε, πολλές φορές οι, οι πολιτικοί στο εσωτερικό των χωρών θεωρούν ότι είναι και επιβάρυνση η ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ισχύει αυτό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να, δίνουν, να δείχνουν την προτιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς, την, προς τους πολίτες τους και χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική ενημέρωση γι' αυτό. Και αυτό πρέπει να αναφέρεται εδώ. Και ένα τελευταίο σημείο κύριε Σιγητά, χτες μιλήσαμε για 105 ε, τροπολογίες που ήρθαν μόνο από τη δική μου την ομάδα για να δούμε πώς, μπορούμε να τις μειώσουμε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε επικοδομητικά. Προσπαθήσαμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις. Οι συμβιβασμοί που, στους οποίους καταλήξαμε μας βοήθησε να μειώσουμε τις τροπολογίες και προσπαθήσαμε με, να επικοινωνήσουμε με τον εισηγητή και χτες καταλήξαμε σε κάποια βασικά θεμελιώδη σημεία. Βρήκαμε εναλλακτικέ λύσεις ή συγχωνεύσαμε κάποιες τροπολογίες και Παρακαλώ απλώς ε, να μας, αποστείλετε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε χτες, ε, ε, εκπονήσαμε χτες. Αυτοί οι, δύο, αυτοί οι συμβασμοί πρέπει να υπάρχουν, ε, να τις έχουν οι ομάδες, οπότε θα θέλαμε να μας τις αποστείλετε γιατί σε κάποιες ε, περιπτώσεις ήταν απλώ μια διαφορά στη διατύπωση, σε κάποιες άλλες ε, περιπτώσεις ο εισηγητή δέχτηκε τι απόψεις μας, οπότε παρακαλώ αυτά που έχετε δεχτεί κύριε εισηγητά να μας τα αποστείλετε έτσι ώστε και οι ομάδε να ξέρουν, να μπορούν να το συζητήσουν, αλλά εγώ εμένω σε αυτά που συμφωνήσαμε χθε. Okay, well, thank you very much. Σας ευχαριστώ και νομίζω μιλώντας ως σκιώδης ότι θα πρέπει να έχουμε όλες τις προτάσεις συμβιβασμού για να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση. Θα ήθελα να κλείσω τη συζήτηση. Κυρία Γκέπχαρτ, θέλετε να επανέλθετε. Μία φράση μόνο, Πρόεδρε. Γιατί θέλω κάτι να προσθέσω. έτσι να αλλάξουμε λιγάκι και διάθεση. Δεν ήξερα ότι οι, οι, επιχειρήσεις και οι μάνατζερ δεν είναι πολίτες. Ό,τι κάνουμε είναι για τους πολίτες. Ε, θα υπάρξει και μία πράξη καινοτομίας, η οποία θα είναι υπέρ των πολιτών επίσης. Κυρία Μπράμπτα. Μπορώ να σας ε, δώσω την ευκαιρία να λάβετε το λόγο. Θέλετε να σχολιάσετε από πλευράς ε, δικής σας προοπτικής και κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω όπως και την τελευταία φορά ότι ε, συμμεριζόμαστε τη διάγνωση που, και την άποψη του εισηγητή δεν είναι αυτός σκοπός η εσωτερική αγορά. Πρέπει να εξυπηρετεί τον Ευρωπαίο πολίτη. Επίσης θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ε, αυτές που ωφελούνται, ίσως όχι ακόμα όσο θα έπρεπε, αλλά θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Και στο έργο που κάνουμε αυτή τη στιγμή για την εσωτερική αγορά, εμείς βλέπουμε την πτυχή που έχει να κάνει με τα ωφέλη που έχουν από τη μια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από την άλλη οι πολίτες. Κάνουμε συστηματική ανάλυση, κάτι που μας λείπει προς το παρόν, για να μπορέσουμε να αποφαρθούμε τι είναι πιο θετικό για την εσωτερική αγορά. Συμφωνούμε λοιπόν με την προσέγγιση που έχει να κάνει με το δούμε ότι από τη μια υπάρχουν οι πολίτε οι οποίοι έχουν ενδεχομένω επιφυλάξει για την εσωτερική αγορά και το πώ ακριβώ λειτουργεί αυτή. Επίσης, η στατιστική έτσι, προσέγγιση να δούμε πώ ακριβώ έχει κατάσταση και να το λάβουμε αυτό υπόψη μα στι αναλύσεις που κάνουμε. Να δούμε τα μέσα για την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλέ τροπολογίε και δι της κυρία Ιβανόβα για τον τρόπο που όταν έχουμε μια παράβαση, κάποια σοβαρή παράβαση, να μπορέσει κανείς γρήγορα να δράσει ε, και την προσφυγή στη δικαιοσύνη όταν δεν έχουμε εφαρμογή οδηγιών. Θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε και σε άλλα σημεία αυτό ενδεχομένω. Επίσης είμαστε θετικοί όσον αφορά το δεχόμενο μιας πράξης για την εσωτερική αγορά και την ε, ιδέα για να υπάρξει μια χάρτα των πολιτών μας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σε αυτή η ιδέα. Και φυσικά όλες τις ιδέες θα τις λάβουμε υπόψη μας στην ανακοίνωση την οποία προετοιμάζει η Επιτροπή και την οποία θα παρουσιάσει στο ε, Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον ε, Ιούνιο. Ευχαριστώ. από πλευράς Κομισιόν για την έκθεση του Λουί και ελπίζω να τύχει υποστήριξη πρόταση. Δίνω το λόγο στο Λουίκ Γκρέκ να μας εξηγήσει πώς θα φτάσει στους συμβιβασμούς και πώς θα τους ε, υφάνει στον κύριο ιστό της έκθεσης. οι σκιώδεις κάναν ό,τι μπορούσαν για να συνεισφέρουν στην έκθεση και θα φτάσουμε στους κατάλληλους συμβιβασμούς. Μετά όμω από τη, τη συζήτηση η ζωή μου γίνεται πιο δύσκολη από μία ώρα πριν. Νομίζω ότι υπήρχε πρόβλημα στα γαλλικά και στα μαλτέζικα, αλλά θα έχετε τις ε, ε μεταφράσει σε τρεις εβδομάδες. Θέλουμε μία ισορροπία και οι κύριοι Κάρας και Γκέπχαρτ είπαν ότι θέλουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία να είναι στα μέτρα του καταναλωτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ε, αδύναμη προσέγγιση. Μία εξορροπημένη προσέγγιση πρέπει να είναι και δυνατή. Άρα η αναζωογόνηση της αγοράς θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Άρα πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Θα κάνω και ορισμένες ε, προφορικές τροπολογίες και μέχρι τις 6 θα έχετε την έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, I'd like to, um, to thank θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λουί Γκρέγ και ευχαριστώ και όλους τους σκιώδεις και από ό,τι φαίνεται η γερμανική και η γαλλική μετάφραση θα είναι διαθέσιμη το απόγευμα. Τα μαλτέζικα είναι πιο δύσκολα. Λυπάμαι, Λουί. Αναμένουμε την ψηφοφορία αύριο. Οι σκιώδεις θα είναι πολύ δραστήριοι και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να επηρεάσουμε με αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ε, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια νέα έκθεση για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και χαίρομαι που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Τέιμιεν Αμπάντ. Είναι η πρώτη σας έκθεση. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Έχουμε Κάμπος Σμιτ. Από την ΚΟΕ e, ο κύριος Σμιτ. Θα ακούσουμε από τον εισηγητή και του Σκιώδης και μετά η Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Και θα δώσω το λόγο και στην κυρία Κολτρέρα από την Επιτροπή. Κύριε Μπάντε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όντω είναι η πρώτη μου έκθεση σε αυτήν την Επιτροπή. Ε, ε, έχω κάνει στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά όχι για αυτό. Τι εδώ. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με αυτέ τι υπηρεσίε γενικού ενδιαφέροντο, Έχει ένα θέμα το οποίο έχει γίνει, είναι μείζωνα σημασία πολιτική. Το είδε και το Συμβούλιο τη Ευρώπη στη Νίκαια. Πέρασε από την οδηγία για τι υπηρεσίε και έχουμε να κάνουμε το πρωτόκολλο των ε, θέμα γενικού συμφέροντος και όλοι, όλοι, μα όλοι διαπιστώνουν ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και όπως ξέρετε η συνθήκη της Λισαβόνας έχει θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτοκόλλο το οποίο δίνει έμφαση σημασία αυτού του θέματος και ε, νομική βάση πάνω σε αυτό. Έχουμε δύο πτυχές. Από τη μια είναι η νομική και από την άλλη η πολιτική. Νομική τώρα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι παρόλες την πρόοδο που έγινε από τη Λισαβόνα και μετά, υπάρχει παρόλα αυτά υπάρχει μια ανασφάλεια όσον αφορά τις νομικές πτυχές. Όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, γιατί από τη μια έχουμε τους κανόνες της ε, αγοράς και από την άλλη τα θέματα που έχουν να κάνουν με ρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις και εδώ έχουμε να κάνουμε τη θέληση αυτή τη εκθεσής, δηλαδή να συμβάλλουμε στο να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε και να ε, προστατεύσουμε και νομικά αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς είμαστε εδώ για να εξετάσουμε ε, διάφορα προβλήματα, ενδεχομένως να δώσουμε απαντήσεις και φυσικά να αξιολογήσουμε τα ενδεχόμενα μέσα που μπορούμε να έχουμε στη θέση μας για να δώσουμε μια εγγύηση όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, εφιστώ την προσοχή στο ότι όχι, να μην περιοριστούμε μόνο στην ε, ε, νομική οπτική γωνία, θα πρέπει να δούμε και την πολιτική διάσταση. Διότι αυτές εδώ οι υπηρεσίες είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν φερρυπίν με παιδικούς σταθμούς, ε, περίθαλψη προστασία ηλικιωμένων, επαγγελματική ε, απασχόληση, όλα αυτά τα θέματα δηλαδή καθημερινής, της καθημερινής ζωής. Και γι' αυτό χρειάζονται λοιπόν μέτρα συγκεκριμένα. Γι' αυτό όταν μιλάμε λοιπόν για αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να καταλάβουμε για ποια πράγματα μιλάμε. Έχει γίνει μια πρόεδρος, ε, πρόοδος στα πλαίσια της Γαλλικής Προεδρίας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα παραπέρα. Έχουμε την εφαρμογή της συνθήκης της Σαββόνας. Όπως σας είπα, ε, έτσι αναγνωρίζεται η σημασία αυτών των υπηρεσιών. Και έτσι περνάμε σε μια νέα ε, δέσμευση της Ευρώπης όπου βλέπουμε την πολιτική διάσταση του θέματος. Αρκεί η μέχρι τώρα εφαρμογή ε, της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής, της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται το θέμα των υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος και στην κρίση που βλέπουμε σήμερα διαπιστώνουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα κινητήρα πρόοδου και εξέλιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι μιλάμε συχνά για μια κοινωνική πολιτική στην αγορά, αλλά έχουμε προβλήματα στην πράξη να περάσουμε. Το κεντρικό θέμα είναι ποια προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά αυτές εδώ τις υπηρεσίες και ποιο είναι το επίπεδο ε, ποιότητας που πρέπει να πετύχουμε. Δηλαδή από τη μια έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση, ένα ε, μέσο πλαίσιο και μετά να το δούμε τομεακά. Κάτι το οποίο αναπτύσσεται σήμερα ή να χρησιμοποιήσουμε το status quo, δηλαδή τη υπάρχουσα ε, οδηγία σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σήμερα έχουμε μια οριζόντια ε, προσέγγιση και μια ε, κάθετη όσον αφορά να δει κανείς τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα. Στόχος δηλαδή να πετύχει κανείς μια αναπάντρεμα αυτών των δύο προσεγγίσεων. Απ' την άλλη, σαν εισήγηση, θα ήθελα να πω να δούμε και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Όπως ξέρετε, αυτές εδώ οι υπηρεσίες ε, είναι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται και σε περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε μέχρι πού θέλουμε να πάμε όσον αφορά την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η συνθήκη της Λατσαβόνας σημειώνει την έμφαση που πρέπει να δοθεί σε εθνικό επίπεδο ούτως ώστε αυτές οι δύο υπηρεσίες να προωθηθούν σε όλη την επικράτεια. Έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, νομικά ή όχι, θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας γιατί καμιά φορά λέμε στα γαλλικά, ξέρετε ότι ε, το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να περάσουμε σε μια ρεαλιστική πολιτική της αγοράς. Αυτά σαν εισήγηση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και εγώ είμαι εδώ πέρα για να ακούσω, να σας ακούσω συνάδελφοι και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Δεν κατέστησα σαφές ότι γνωμοδοτείτε έναντι μιας έκθεσης Επιτροπής Απασχόλησης, η οποία ασχολείται με τη γενικότερη εμβέλεια του θέματος. Μπορείτε να μας πείτε πώς έχει η κατάσταση στην Επιτροπή Απασχόλησης πριν μιλήσουν οι σκιώδεις. Μάλιστα. Στην Επιτροπή Απασχόλησης τα πράγματα είναι στο μηδέν. Ε, οι συζητάνε. Εγώ είμαι σε επαφή με τον εισηγητή και είμαστε σε μια φάση όπου υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις όπου δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο ε, στοιχείο. Ελπίζω όμως σύντομα να έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά το θέμα που αφορά τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ωραία. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε έτσι και εμείς να καθοδηγήσουμε με τις δικές μας πράξεις αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ακούσουμε τώρα τους Κιώδης. Ο κύριος Κοραγία Δεκάμπος καταρχήν. Ευχαριστώ θα ήθελα να τονίσω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπε ο εισηγητής και θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σε ορισμένα σημεία που αποτελούν το ιστορικό αυτής της συζήτησης οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ανέκυψαν από την αλληλεγγύη, από την κοινωνική ιστορία αλληλεγγύης, όχι από την ιστορία της αγοράς. Αργότερα φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν κακό να εισαγάγουμε στοιχεία απόδοσης της αγοράς για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα αυτές τις υπηρεσίες. Εάν όμως ήταν αντίθετη πορεία της ιστορίας τότε. Εάν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν ανακύψει από τους μηχανισμούς της αγοράς, τότε θα είχαμε μία πιο αδική ιστορία. Στη χώρα μου, εκτός από τις συντάξεις το, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας δημιουργήθηκε εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν υπήρχε το ΕΣΥ, θα υπήρχαν οι υπηρεσίες υγείας ε, καλής ποιότητας, αλλά και πολύ κακής για, τις, ε, ε, για τους πολίτες ενδοχώρας. Όπως είπε ο εισηγητής, υπάρχουν νομικά ζητήματα και οικονομικά θέματα που δεν έχουν επιληθεί. Διότι οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να ισχύει για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Διότι υπάρχει έλλειμμα στην αγορά και χρειάζεται νέα επαναρρύθμιση της αγοράς. θα πρέπει να προβάλλουμε τρεις αξίες σε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, την ποιότητα, την αποδοτικότητα, αλλά υπάρχει και μία άλλη αξία που είναι η αρχή της ισονομίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Εάν δεν υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ των ε, τριών ε, πτυχών, τότε δεν υπάρχει αποδοτικότητα διότι πολλές φορές υπάρχουν αντιφατικά σχήματα μεταξύ ισονομίας και δικαιοσύνης. Γι' αυτό θα πρέπει να φτάσουμε σε μία επανεξισορρόπηση. Βεβαίως η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει την σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος, γι' αυτό επανεκκίνησε και αυτή η συζήτηση. Θα πρέπει να εξεύρουμε και τα κατάλληλα νομικά μέσα και νομοθετικά πλαίσια, όπως ανέκυψαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Γι' αυτό πάντα μιλάμε και για την εταιρικότητα δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Το θέμα της επικουρικότητας πώς έχει. Το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι ε, θέμα στο οποίο θα προσφύγουμε σε τελευταία ανάλυση. Δεν μπορεί κάθε χώρα να λέει ότι αυτό είναι ένα θέμα επικουρικότητας και δεν επιτρέπω στους κοινοτικούς ε, μηχανισμούς να μπουν στην, ε, στις δικές μας κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται όμως να προσφύγουμε σε αυτό το τελευταίο προμαχώνα. Εάν ε, δεχτούμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου του 2006 για, την, ε, για τις Common Values and Principles στον ε, τομέα της υγείας, γιατί τότε συζητούσαμε κατά πόσο ο τομέας υγείας θα ενταχθεί στην οδηγία περί και αυτή η συζήτηση διασάφησε πολλά πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή θα πρέπει να είναι και η βάση που να διέπει τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναρκοπέδιο. Πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπε ο και ελπίζω όντως να επιτύχει, να μην πατήσει καμιά νάρκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει όντω να δούμε αυτού τους ε, τομεί που θεωρούνται οριζόντι σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα και στους οποίους κατά μεγάλο βαθμό έχουμε αποτύχει. Όλοι θυμόμαστε την κινητικότητα των ασθενών και τα δικαιώματά τους και τη συζήτηση που είχε γίνει. Καλό για την αγορά καλό και για τους ασθενεί. Μπλοκαρίστηκε. Και ακόμη μπλοκαρισμένο είναι. Και δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά ως κοινοβούλιο για να παράσχουμε αυτού του είδους την πρόνοια και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς, τους πολίτες της Ευρώπης οι ρίζε λέει δεν είναι στην αγορά. Εγώ είμαι από τον Βορρά, από ένα μικρό χωριό. Οι ρίζε πάντα βρίσκονταν στην οικογένεια. Η οικογένεια τα αναλάμβανε τα θέματα αυτά. Η φτώχεια, η φροντίδα των ηλικιωμένων, τα παιδιά, όλα τα ρύθμιζε η οικογένεια. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Και τώρα το κράτος και το τοπικό και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση αναλαμβάνουν αυτό το χρέος. Και οι φόροι και οι, οι πληρωμές μάλλον γίνονται μέσω της φορολογίας. Ε, αυτά έχει η επικουρικότητα. Μάλκομ, τι θα έλεγες εσύ να μην υπάρχει, τι λέτε στη Βρετανία, να μην υπάρχει φορολόγηση χωρίς να υπάρχει εκπροσώπηση. Ε, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιους βασικούς κανόνες στην Ευρώπη. Σε πολλούς τομείς το προσπαθούμε, υπόθηκε ήδη. Διαχείριση αποβλήτων ας πούμε, στη δική μου τη χώρα. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν έχουν εφαρμόσει την ευρωπαϊκή οδηγία, όχι τη θεωρούν, καλύτερα τα καταφέρνουν μόνοι τους μας λένε, κάνουν δημόσιες προμήθειες και ε, βρίσκονται λίγο στο περιθώριο. Αλλά εντάξει, δεν του πειράζει. Αυτοί έχουν βρει τρόπο να τα λύνουν μόνο του το πρόβλημα. Και για άλλου πιο περίπλοκου τομεί το ίδιο. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτό το πρωτόκολλο με σωστό τρόπο, παρόλο που Θεωρώ ότι πολλοί από τους συναδέλφους πιστεύουν ότι αν θέλουμε να έχουμε πιο σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μας αρέσει λίγο παραπάνω από όσο μας αρέσει τώρα, ε, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιες κοινωνικές πτυχές και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Νομίζω όμως ότι αυτή είναι η λάθος μέθοδος, ο λάθος τρόπος, τουλάχιστον για τη δική μου τη χώρα. πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, εμείς τουλάχιστον θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, γιατί πιστεύουμε ότι μία κοινότητα, μία τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει κάποιους κανόνες που αφορούν την, τα σχολεία, την προορία για τα παιδιά, την φροντίδα των ηλικιωμένων, την υγεία. Εντάξει, πρέπει φυσικά να υπάρχει και ένα ελάχιστο όριο, αλλά αν θέλετε να περάσουμε σε μία κοινότητα όπου δαπανούμε τα περισσότερα κονδύλια για τους ηλικιωμένους, Εντάξει, α το κάνουμε, αλλά θα αυξηθούν και οι φόροι. Να το ξέρετε αυτό. Στη δική μου τη χώρα πληρώνουμε 32% τοπικούς φόρους, τοπικούς και περιφερειακούς. Επομένως, μπορεί κανείς να διαλέξει τι είδους υπηρεσίες προτιμά. Οπότε, αν λέμε ότι πρέπει να έχουμε κάποιους κοινούς κανόνες ή τέλος πάντων ένα μια ισορροπία δυνάμεων. Εντάξει, αυτό καλό είναι. Αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα για να εξευρεθεί μια ισόρροπη προσέγγιση. Εγώ διάβασα κάποια από τα έγγραφα της Κομισιόν για το πώς προτείνει η Κομισιόν να προχωρήσουμε. Και αυτοί λένε να προχωρήσουμε προσεκτικά. Για να κλείσω, λοιπόν, Πρόεδρε, εγώ ευχαρίστω να ακούσω όλα τα επιχειρήματα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε καταρχήν με τα οριζόντια θέματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει αρκετά. Τουλάχιστον η δική μου άποψη αυτή είναι. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι μεγάλες αρχές που έδειξε ο κύριος Σαμπάντ μου φαίνονται πολύ σωστές και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος έλεγα. Απ' την άλλη θα ήθελα να πω σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος Ούλε Σμιτ ε, διαφωνώ διότι δεν θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στι θέματα που έχουν να κάνουν με διασυνοριακής φύσεω ε, πτυχέ, αλλά θέλουμε να δούμε πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς στην επικράτειά του υψηλέ υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Όχι να πάει δηλαδή σε μια άλλη χώρα για να έχει όφελος αυτών των υπηρεσιών, έχοντας δηλαδή διαφορετικά μοντέλα σε κάθε χώρα. Το θέμα είναι, ο στόχος μας είναι η, το επίπεδο και η ποιότητα. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί κατά τη διάρκεια που έγινε η εκστρατεία για να γίνει η επανεκλογή της. Είχαμε τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος είχε υποσχεθεί ένα επίπεδο ποιότητας όσον αφορά ε, τις υπηρεσίες αυτές σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχει κανείς με τις υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να προχωρήσουμε και είναι σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει την πρωτοβουλία και να τα φέρει επιτάπητος. Επίσης, να πω... Ε, δεν ξέρω αν έχει κάνει ήδη επαφές ο εισηγητής της Επιτροπής μας με τις ε, ομάδες με την ομάδα μάλλον για τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Ε, είμαστε από όλες τις ομάδες εκπροσωπημένοι εκεί πέρα, σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και μαζί με την Επιτροπή να προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα περιεχόμενο στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών όπως είχε, το είχε προτείνει και ο πρόεδρος της Επιτροπής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την οικοδόμηση αυτού του έργου. Απ' την άλλη, αυτές εδώ οι υπηρεσίες είναι και οι υπηρεσίες που έχουν την οικονομική τους διάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν να κάνουν και με την αξιολόγηση της Επιτροπής. Υπάρχει το θέμα του το, το γνωστό πακέτο Monty Cross και θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα σχετιστεί το όλο θέμα με την αξιολόγηση. και να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, ποιες ε, κριτικές έχουν γίνει ενδεχομένως από τους διαφόρους εταίρους, ποιες είναι οι θέσεις που θα πρέπει και οι αντιδράσεις ε, που θα πρέπει να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες οι αντιδράσεις του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίλαν δεν είναι εδώ. Θα συνεισφέρουμε και εμείς Άρα η κυρία Βανιούρο έχει το λόγο. Αντιπρόεδρος και μετά θα σχολιάσει η Επιτροπή πριν συνοψίσει ο κύριος Σαμπάντ. Ευχαριστώ. Σύντομα να πω στον κύριο Αμπάντ ότι πραγματικά έθεσε τα σωστά ερωτήματα, τον συγχαίρω. Θα έχουμε μια, ένα σωστό διάλογο, τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Είναι θεμελιώδος. Και όπως είπε και ο Αντώνιο, είναι σημαντικό για τους πολίτες. Τώρα, μιλάτε για το αν το μέσο της συνθήκης ε, Λισαβόνας είναι αρκετό. Εγώ θα έλεγα όχι. Ξέρετε, ένα μέσο έχει να κάνει με το πώς ακριβώς το χρησιμοποιεί κανείς, με ποιο στόχο. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του μέσου που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλοι εξάλλου συμφωνούμε Είμαστε σε μια κρίση οικονομική, κοινωνική που δεν έχουμε ξαναδεί. Και πραγματικά υπάρχουν εδώ οι πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη ε, υπηρεσιών στην καθημερινή τους ζωή. Υπάρχουν άτομα τα οποία βρίσκονται σε ε, δύσκολη κατάσταση. Και έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα και με την οικονομική πτυχή, δηλαδή με θέσει εργασίες οι οποίε δεν γίνεται να, ξέρετε, να μεταφερθούν κάπου αλλού όπω γίνεται με τι επιχειρήσει. Θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε ποια προσέγγιση, ποιο είδους προσέγγιση θα έχουμε. Και το τρίτο θέμα που είπατε για την, την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ανησυχούμε όντως όσον αφορά την αξιολόγηση αυτής της ε, ε, και αναρωτιόμαστε πώ θα περάσει η εφαρμογή της στις χώρες μέλη. Υπάρχει ένας τομέα, μια γκρίζα ζώνη εδώ. Θα έχουμε λοιπόν διάλογο εδώ, αλλά και σε άλλες επιτροπέ. Τι θα έχουμε, μια οδηγία πλαίσιο ή οδηγίες ε, ε, τομεακά θα λέγαμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το θέμα είναι τώρα μια προσέγγιση οριζόντια ή κάθετη. Εγώ θα πρότεινα περισσότερο ότι όχι μόνο να πούμε οριζόντια ή κάθετη προσέγγιση, αλλά μια σφαιρική. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει κάτι το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο για τις, για τις δημόσιες προμήθειες. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε με πάρα πολλά θέματα. Έχουμε να κάνουμε με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, τη φροντίδα των παιδιών, ε, εργατικές κατοικίες, το περιβάλλον. Όλα αυτά θα πρέπει ε, να τα έχουμε υπόψη. Νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δούμε τους διάφορους επιμέρους τομείς για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σωστό προβληματισμό γιατί το είπε και ο Αντώνιο ότι τα θέματα έχουν να κάνουν τόσο με την ε, ε, αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την προσέγγιση ε, στις υπηρεσίες από όλους. Είναι πολύπτυχο, πολύπλευρο το θέμα και θα πρέπει φυσικά στόχος μας να είναι η συνένεση. Ο χρόνος είναι λίγος και οι πολίτες έχουν ανάγκες και υποφέρουν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Κούτραβα νομίζω ότι θα μιλήσει εκ μέρους της Κομισιόν και αν μπορείτε πείτε μας και αυτό το σημείο που υπάρχει στο πρόγραμμα εργασίας για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και για το ποιοτικό πλαίσιο. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για το πώς βλέπει η Κομισιόν την όλη κατάσταση. Ευχαριστώ. Να σας πω ποια είναι η προσέγγιση της Κομισιόν για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και θα αναφερθώ στα σημεία αυτά που βρίσκονται στο πρόγραμμα εργασίας. Καταρχήν να πω ότι συμμεριζόμαστε τις ε, απόψεις των ε, διαφόρων ομιλητών για την σημασία των, οικονομικών επιχειρη... των κοινωνικών επιχειρη... Ε, ε, υπηρεσιών συγγνώμη, στην, στην κοινωνία μας, ώστε να είναι η κοινωνία πιο συνεκτική και αποτελούν το εφαλτήριο για τέτοιου είδους κρίσεις. Όπως αυτή που περνούμε τώρα. Η Κομισιόν στη διετή έκθεσή της από το 2008 αναφέρει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι κρίσιμη πηγή παροχής θέσεων εργασίας. Οπότε για όλου αυτούς τους λόγους η Κομισιόν πάντα έδινε ιδιαίτερη σημασία στις κοινωνικές υπηρεσίες. Καταρχήν να αναφερθώ στο γιατί αυτές οι υπηρεσίες, των οποίων η χρηματοδότηση και η οργανώση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων των ευρωπαϊκών την τελευταία δεκαετία έχουν υπάρξει διάφορες διαδικασίες αναθεώρησης, ε, μεταρρύθμισης στα κράτη-μέλη, που δεν, ε, των οποίων δεν ηγείται η Κομισιόν. Είχαν διάφορες μορφές, όλες όμως έδειχναν την ίδια τάση. Μία από τις τάσεις αυτές ήταν η εξωτερήκευση. Η ανάληψη δηλαδή τη παροχή υπηρεσιών από μη κερδοφόρου ή από ε, ή κυβερνητικού οργανισμού. εμπίπτουν βέβαια και στους κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Οι υπηρεσίες που, που, προβλέπονται από, που προφέρονται από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι ε, υποκειμενικές, ενώ αυτές που προσφέρονται από το κράτος δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οικονομική δραστηριότητα χωριστή. Η Άξις λοιπόν της ευαισθητοποίησης που εμπίπτει και σε όλη τη διαδικασία των κοινωτικών κανόνων θα πρέπει να διαλευκανθεί. Να σας ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για την εφαρμογή των κανόνων, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για την, για, την ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να οδηγήσει σε απελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών. Αυτό είναι λάθος. Οι ε, αρχές στα κράτη-μέλη μπορούν εφόσον αυτό είναι λογικό και ανάλογο, μπορούν να δώσουν ειδικά δικαιώματα ή αποκλειστική αρμοδιότητα ή να περιορίσουν τους, ε, την παροχή υπηρεσιών σε κάποιους ε, παροχής υπηρεσιών. Άλλη ε, παρεξήγηση, ότι οδηγείται σε απορρίθμιση, οδηγούνται σε απορρίθμιση αυτές οι υπηρεσίες λόγω των κοινωνικών κανόνων. Όχι καθόλου, ελευθερία εγκατάστασης και άλλες διατάξεις ισχύουν εδώ που είναι, είτε είναι απαραίτητες και αναλογικές και έχουν ως στόχο να προωθήσουν το κοινό συμφέρον. Οι γενικοί στόχοι λοιπόν λαμβάνονται υπόψη για τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, μια άλλη παρεξήγηση. Ιδιωτικοποίηση. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει να γίνουν ιδιωτικοποίησεις. Καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ρυθμίσει ε, την, ε, την, μέσω των, ε, να ρυθμίσει την, τις υπηρεσίες αυτές μέσω όμως των κανόνων που θέτουν τα κράτη-μέλη, οι, οι δημόσιες αρχές. Επίσης, όταν οι δημόσιες αρχές πρέπει να, να εφαρμόσουν ε, κανόνες δημοσίων προμηθειών, μπορούν να, να ε, θέσουν ε, προϋποθέσεις ποιότητας, έτσι ώστε να πληρούνται κάποια κριτήρια, κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες περιβαλλοντικές ακόμη προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τώρα, σύντομα να πω ότι οι υπάρχοντες κανόνες λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαιτερότητες τον, ε, του τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Κάποιοι από εσά μιλήσατε για το παλιό πακέτο Μόντε Monte Cruz και για τη χρηματοδότηση. Ούτως ή άλλως όμως αυτές, ε, αυτό εμπίπτει στις, ε, κρατικούς κανόνες. Στην έκθεση από το 2008 το αναφέρουμε ήδη ότι 90% κατά μέσο όρο, 90% του κόστου των κοινωνικών υπηρεσιών καλύπτεται από το δημόσιο τομέα. Και η ε, οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες δίνει επίσης ε, ειδικό ρόλο στις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι, οι... Κάποιες ε, κοινωνικές υπηρεσίες αναφέρονται στο παράρτημα 2β είναι ιδεατή η κατάσταση αυτή? Όχι, καθόλου, καθόλου. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν κολλήματα και αυτά ακριβώς τα κολλήματα και τις δυσκολίες η Κομισιόν προσπαθεί να τα επιλύσει. Από το 2007 έχει δώσει έγγραφα με, συχνά, ε, με συχνές ερωτήσεις που συνδέονται και που έχουμε λάβει από του stakeholders, από του διάφορου εμπλεκόμένου ειδικά για τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Και έχουμε δώσει λειτουργικέ απαντήσει. Επίση, έχουμε ένα διαλειτουργικό, μια διαλειτουργική, πύλη ενημέρωση για να, ενημερώνονται, να ενημερώνονται και οι δημόσιε αρχέ για τι κοινωνικέ υπηρεσίε και όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Και επίση το 2009 ξεκινήσαμε μια μια πρωτοβουλία κατάρτισης για τι τοπικέ και τι περιφερειακέ αρχέ. Ε, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα ε, τους κανόνες. Παρόλο που έχουμε κάποιες αμφιβολίες για τα γενικά μέσα, το... για τις κοινωνικές ε, υπηρεσίες, δεν αποκλείουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες που μπορεί να χρειάζονται τροποποίηση. Uh, Βεβαίως όλα αυτά υπόκειται πάντα σε αξιολόγηση η Κομισιόν είναι πραγματικά πολύ ενεργή στην, ε, στον τομέα αυτό. Έχει δημιουργήσει μία ε, ομάδα εργασία ε, με την Επιτροπή Κοινωνική Προστασία και εκεί έχουν καταδειχθεί κάποιε κάποιες κάποιοι τομεί που χρειάζονται περαιτέρω προσοχή. Ας πούμε οι κανόνες για τι για τις δημόσιες προμήθειες, πιθανές κανόνε τους αυτούς για κάποιε έκτακτες περιπτώσει και για παροχή υπηρεσιών από μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους ενδιαφερόμενου, έτσι ώστε να δούμε ποιε είναι οι προτάσεις τους. Πάμε στην ε, ανακοίνωση που έγινε με το πρόγραμμα εργασίας. Όντω. ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση για το ποιοτικό ε, πλαίσιο για τις οικονομικές υπηρεσίες, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας γενικώ, αλλά για τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος εξεκολουθούμε να ε, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης ενός ειδικού πλαισίου ποιότητας. Υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία επίσης ε, ασχολείται με το θέμα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα του τρίτου φόρουμ που οργανώνει η Βελγική Προεδρία με την Κομισιόν. ο οποίος ακολουθεί την σύσταση που έχει στείλει το Κοινοβούλιο. Οι άλλες δύο πρωτοβουλίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασίας αφορούν το πακέτο Altmark, την αξιολόγηση του πακέτου και ίσως και την αναθεώρησή του. Ελπίζω να κάλυψα τις απορίες σας, βεβαίως αν υπάρχουν κι άλλες, εδώ είμαι. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούτρα. Ήσασταν απόλυτα σαφής, μα απόλυτα, ιδιαίτερα για το ρόλο αυτής της Επιτροπής, κάτι το οποίο θα λάβει υπόψη ο εισηγητής. Δίνω το λόγο στον κύριο Αμπάντ λοιπόν για να μας ε, μιλήσει για τα επόμενα βήματα. Έχουμε ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα εδώ αλλά εξαρτάται από τις συζητήσεις του με την Επιτροπή Απασχόλησης για να δούμε πού θα εστιάσουμε την προσοχή μας, διότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικό το να ε, συντάξουμε μια έκθεση τη στιγμή που η Επιτροπή Απασχόλησης δεν έχει συμφωνήσει για το πεδίο εμβέλεια. Μάλιστα, ευχαριστώ. Να Ευχαριστώ και όλους τους προλαλήσαντες που εμπλουτίζουν αυτή την έκθεση και τη Σκιώδη εισηγήτρια. Όσον αφορά τώρα για το ερώτημα που θέσατε, όσον αφορά την αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή Απασχόλησης, το θέμα είναι αν θα πρέπει να γίνει μια έκθεση πρωτοβουλίας νομοθετικής φύσεως ή όχι. Σύμφωνα με το αίτημα της Σοσιαλιστικής Ομάδας μου δώσα μια προθεσμία της 20 Μαΐου με το διάλογο που έχουμε εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο. Άκουσα και από την Επιτροπή ε, που αναφέρθηκε στο θέμα που αφορά το περιεχόμενο και τις διευκρινήσεις του περιεχομένου ε, είναι σαφές ότι οι υπηρεσίες για τις οποίες συζητάμε εδώ είναι σημαντικές για να πετύχουμε μια κοινωνική ε, συνοχή. Υπηρεσίες στις οποίες όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση. Νομίζω η προσέγγιση ε, πρέπει να είναι σφαιρική και είμαι έτοιμο να συνεργαστώ με την ομάδα η οποία δουλεύει για τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος και είναι σαφές ότι όλο αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε στα πλαίσια της σημερινής κρίσης, της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν αυτές οι υπηρεσίες όσον αφορά την απασχόληση. Έχουμε και το θέμα των ε, κρατικών επιδοτήσεων, ε, διασυνοριακής φύσεως πτυχές Ε, που δεν είναι άμεσα φυσικά το θέμα της εκθέσεως. Θα πρέπει όμως να δούμε όλα αυτά εδώ τα θέματα και επιμένω η προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε να είναι ρεαλιστική. Ευχαριστώ. Okay, well, uh, Προτείνω να το εντάξουμε στην ημερήσια διάταξη το θέμα όταν ε, έχετε προχωρήσει και μπορούμε να το συσχετίσουμε με το τι κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης. Αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να δούμε τις δραστηριότητες της Επιτροπής σε αυτό το τομέα και να δούμε ποια είναι, ποια είναι η πραγματική συνεισφορά αυτής της Επιτροπής υπό μορφή προστιθέμενης αξίας. Εάν η Επιτροπή Απασχόλησης ε, προτείνει μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τότε θα έχουμε επιμερισμένη αρμοδιότητα και θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία μαζί τους. Μπορούμε να το αφήσουμε λοιπόν αυτό σε εσάς και θα πρέπει να δούμε πώς ορισμένες πτυχές της τυποποίησης μπορεί να επηρεάσουν το θέμα των ε, προτύπων ποιότητας. Γιατί η τυποποίηση έχει σχέση και με τις υπηρεσίες, ε, καθώς και με τα αγαθά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι το σχέδιο γνωμοδότησης Fox σε συσχετισμό με την Επιτροπή Γεωργίας. Κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για το δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες και την βελτίωση της λειτουργίας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του Σκιώδης και την ε, Γραμματεία γιατί με βοήθησαν. Ή έλαβα πολλά επικοδομητικά σχόλια και προσπάθησα να τα εντάξω στη γνωμοδότηση. Ο κύριος Ζουδέ έκανε, ανέφερε πολλά σημεία που βελτιώνουν τη διαφάνεια στην αλυσίδα και καλύτερη ενσυνειδητότητα των ε, δικαιωμάτων των ε, συμβατικών δικαιωμάτων σε σχέση με τις συγκεκριμένες πρακτικές. Συμφωνώ με την κυρία Βέστφαλ ότι οι συμβατικές σχέσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε πιο ασφαλές έδαφος και ζήτησα να ε, ζητηθεί η σύνταξη τέτοιων συμβάσεων στα πλαίσια της ε, αλυσίδας διατροφής, αλλά δεν θα ήταν έμπρακτα σωστό όλα αυτά να γίνουν γραπτός. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να άρουμε τις αθέμητες πρακτικές έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι αθέμητες πρακτικές ε, έμπρακτα διότι θα ήταν επιζήμιες ε, και για τον καταναλωτή. Ο κύριος Λάιν είπε ότι η ανισορροπία δεν έγκυται στο οικονομικό μέγεθος των φορέων, αλλά και στην αγοραία δύναμη που έχουν στη διάθεσή τους. Συμφωνώ με τα λεγόμενα του και πιστεύω ότι εάν υπάρχει ισορροπία θα λειτουργήσει καλύτερα και η διατροφική αλυσίδα και αυτά υπέρ του καταναλωτή. Επίσης, η Επιτροπή Υψηλού Επίπεδου ασχολήθηκε με την ανταγωνιστικότητα της αγροτροφικής αλυσίδας, αγροδιατροφικής αλυσίδας, για να άρουμε τις ανισορροπίες στα πλαίσια της διατροφικής αλυσίδας. Θα ήθελα να συνεργαστώ με τους άλλους σκιώδεις για να καλύψω και θέματα που δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και θα συντάξω και τροπολογίες έτσι ώστε και οι προμηθευτές να οργανωθούν κατά τρόπο ώστε να αυξήσουν την επιρροή τους και τη δύναμη διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν τις αθέμητες πρακτικές και να προωθήσουν ευκολότερες πρακτικές ενσωμάτωσης και να υπάρχουν σωστές πληροφορίες ως προς τη σήμανση και εποπτεία των τιμών, έτσι ώστε να έχουμε και καλύτερα μέσα σύγκρισης τιμών. Θα ήθελα να λάβω τροπολογίες από τους άλλους σκιώδεις σε σχέση με τα σημεία αυτά. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσουμε και έναντι του κυρίου Μποβέ, δηλαδή της Επιτροπής Γεωργίας. Ευχαριστούμε κύριε Φόξ. Θα ήθελα τώρα οι σκιώδεις να, δώσουν, να λάβουν το λόγο. Ζουβέ. for εγώ θα μιλήσω ε, για τους πράσινους, ίσως και η κυρία Ρούλε και ο κύριος Λοντέρο θα μας πει λίγα λόγια. Θα πρέπει να είμαστε σύντομοι, γιατί έχουμε και μια παρουσίαση στις 12. Ο κύριος Ζουβέ. voyez que nous sommes écoutés. Président, remercier. Merci, Monsieur Monsieur le Président. À moi de remercier Fox pour. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φόξ για την εξαιρετική του εργασία. Θα είμαι σύντομος. Η εργασία αυτή είναι σημαντική για τρεις λόγους, γιατί αφορά τους καταναλωτές. 16% του προϋπολογισμού των οικοκυριών πάει στη διατροφή. Αφορά και τους γεωργούς, διότι όταν οι τιμές κατανάλωσης πέφτουν, τότε πέφτουν και τα γεωργικά εισοδήματα και όταν οι τιμές ε, κατανάλωσης αυξάνουν δεν σημαίνει ότι αυξάνει και το εισόδημα των γεωργών. Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είμαστε αυτάρκης από πλευράς διατροφής. Ίσως φαίνεται κάτι το κεκτημένο και το οριστικό όπως η ειρήνη, που δεν μας απασχολεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι πρόβλημα αλλά ε, ε, όταν γνωρίζουμε κρίση στον τομέα της υγείας και των υγειονομικών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον σημαντικό χαρακτήρα της αυτάρκειας. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Φόξ, αλλά θα ήθελα να πω ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των ε, θυγατρικών έτσι ώστε οι γεωργοί να ε, οργανώνονται σε συνεταιρισμούς παραγωγών για να είναι πιο δυνατοί και να μπορέσουν να έχουν ειδικό βάρος της διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την αλυσίδα παραγωγής. Δεν την γνωρίζουμε επαρκώς και παραδοσιακά υπάρχει κατακραυγή ε, ως προς την ε, αλυσίδα προμήθειας. Αλλά όταν μιλάμε για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ξεχνάμε ορισμένους ε, τομείς που δεν αναγνωρίζουμε σαφώς. Ξέρετε ότι σήμερα 20% των γευμάτων παράγονται από τις βιομηχανίες συλλογικής εστίασης που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ε, οικονομική δυναμική. Θα σταματήσω, λέει ο κύριος ε, Μποβέ. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η αργάνωση των εμπλεκόμενων φορέων και η διαφάνεια των εμπλεκόμενων φορέων και σας μίλησα για τη συλλογική εστίαση η οποία πολλές φορές δεν την χάνει αναγνώριση. Ευχαριστούμε κύριε ε, Ζουβέ, κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Σάλφος είναι ένα ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή, ή συνάδελφος μάλλον, και πρέπει να την αντικαταστήσω εγώ. Ε, να ευχαριστήσει την, ε, τον κύριο Φόξ για τη δουλειά που έκανε και χαιρέται πολύ που ο κύριος Φόξ σαφώς ανέλαβε το εγχείρημα αυτό από την πλευρά της προστασίας της αγοράς και των καταναλωτών. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε επικεντρωθεί στον τομέα αυτό και μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Επίσης, συμφωνεί με αυτή την ε, ε, ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των σούπερ μάρκετ, της αγοράς, των αγροτών, των, ε, των διατροφικών προϊόντων, της διατροφικής αλυσίδας, να την ξανασυζητήσουμε και είναι φυσικά θέμα να υπάρξει ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των φορέων, όπως το είπε και ο συνάδελφος. Επίσης χαιρετίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και για τη δική μας την ομάδα αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο γιατί οι εξαρτήσεις που υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς πρέπει να τις δούμε. Να γίνουν έτσι πιο προφανείς και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν επιφέρουμε διαφάνεια. Βέβαια αυτό δεν είναι αρκετό απάντηση για τα προβλήματα που υπάρχουν και η δική μας ομάδα θα κάνει κάποιες προτάσεις ως προς αυτό, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές. Επίσης η ομάδα μας, κάτι που σίγουρα θα θέσει, με ποιο τρόπο δεν ξέρω ακόμα, είναι το θέμα των ε, συμβάσεων. Λέτε ότι ε, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό ή δεν γίνεται με απόλυτα σωστό ε, τρόπο ε, στον τομέα τη γεωργίας και δεν πρέπει γενικώ να καταργηθεί. Αν δηλαδή δύο γεωργοί θέλουν μεταξύ του να συμφωνήσουν για κάτι, αυτό πρέπει να μπορούν να το, να το κάνουν. Αλλά πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του γεωργού και μια μεγάλη εταιρεία με την οποία αυτό κάνει δουλειέ. Και Νομίζω ότι θα πρέπει να, γίνουν και, να γίνονται και κάποιε γραπτές, κάποια γραπτά συμβόλαια σε τέτοιε περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς μπορούμε να το θέσουμε αυτό στην έκθεση και από ό,τι φαίνεται ε, αναμένονται αρκετέ αντιφατικέ συζητήσει. Ε, εντάξει, αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Επίση, η κυρία Βέσφαλ πιστεύει ότι στα ερωτήματα αυτά, στα θέματα αυτά, Χρειαζόμαστε καλή συνεργασία με τον εισηγητή και χαίρεται πολύ που ο εισηγητής έχει πάντα ευήκον ους για τις υπόλοιπες απόψεις. Είπατε κι εσείς ότι θα θέλετε να υποβάλλετε κάποιες τροπολογίες για να κλείσουν τα κενά και βεβαίως και εμείς αν μπορούμε να συμβάλλουμε. Φυσικά πάντα είναι καλό αυτό αν μπορούμε να συμβάλλουμε ως ομάδα ώστε να σα βοηθήσουμε στο έργο σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σμιτ. Εγώ ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να κάνω τον κύριο Λάιον. Θα είναι δύσκολο. Ζητά συγγνώμη που δεν είναι παρόν σήμερα. είναι στη Βρετανία και κάνει προεκλογική εκστρατεία. ορίζετε την γνωμοδότησή του κυρίου Φόξ για την προσοχή των καταναλωτών. Το Τέσκο, ένα από, τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, έκανε κέρδη 3,17 δισεκατομμύρια λίρες. Αν δεν είναι λίρες θα είναι ευρώ. Πάντως το ποσό παραμένει το ίδιο. 10% αύξηση επίσης στον, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο όταν οι ε, γεωργοί πληρώνονται όλο και λιγότερο και οι, οι ε, καταναλωτές πληρώνουν όλο και περισσότερο. Αυτό δείχνει την μεγάλη ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ των ε, καταναλωτών, των γεωργών, των μεταποιητών και ε, πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι stakeholders ώστε να υπάρξει καλύτερη λειτουργία και πιο δίκαιη αλυσίδα διανομής. Επίσης ε, θεωρεί ότι η έκθεση αντιμετωπίζει το θέμα των ε, αθέμητων συμβασιακών πρακτικών και ο κύριος Λάιον επίσης χαίρεται που ο κύριος Φόξ κάνει αναφορά στον διαμεσολαβητή. Κάτι που ο κύριος Μπουβί δεν ανέφερε στη δική του, στο δικό του σχέδιο έκθεσης. Ο κύριος Λάιον θα υποβάλει δύο τροπολογίες. Μία για τις αφέμητε πρακτικές, ώστε να είναι σαφές ποιες είναι οι καταστροφικές πρακτικές για, για την αλυσίδα διανομής και επίσης ανταγωνιστικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της αλυσίδας διανομής. Τέλο Πρόεδρε, ο κύριο Λάιον θεωρεί ότι οι συζητήσει εδώ θα ενσωματωθούν στην ε, δουλειά που κάνει και η Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη συνέργεια μεταξύ των δύο επιτροπών. Επίση, θα ήθελε να σα καλέσει όλου να παραστείτε σε μια ακρόαση που, κάνει, που οργανώνει η Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων Γεωργίας ε, τον Μάιο. Ακόμα πότε δεν ξέρουμε, αλλά θα ενημερωθείτε εν καιρό. Uh, Ευχαριστώ. Δεν είναι ο μόνος ο κύριος ε, Λάιον που, είναι, που εμπλέκεται στις ε, προεκλογικές εξαδίες, είναι και άλλοι. Η κυρία Ρούλε. Και εγώ είμαι σκιώδης. Θα είμαι σύντομη. Και εγώ χαιρετίζω το γεγονό ότι ο εισηγητή έχει επικεντρωθεί στα σημεία αυτά, τα οποία επεξεργαζόμαστε και εμεί στην Επιτροπή. Ο διαμεσολαβητή είναι σωστό. Στον κύριο, στην έκθεση του κυρίου Μπουβέ δεν αναφέρεται. Νομίζω ότι αυτή είναι κυρίω ε, καθήκον τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ να θέτει τέτοια θέματα, έτσι ώστε να ενισχύει την προστασία των καταναλωτών μέσω και των ενώσεων των καταναλωτών που αποστέλουν τέτοια αιτήματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε ω προ αυτό. Κατά τα λοιπά, ακούστηκαν όλα τα σημαντικά στην έκθεσή σα, αναφέρονται και χαίρομαι που έχουμε μια τέτοια καλή βάση βάση για τη συνεργασία μας, κυρίως με το θέμα αυτό, με, τις, ε, με το δίκαιο συμβάσεων. Äh, και με τις ε, προσθήκες που θα κάνουμε ελπίζουμε να βοηθήσουμε και την ε, Επιτροπή Γεωργίας. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλα μέλη που θέλουν το λόγο, τότε ο κύριος Λοντέρο να κάνει κάποια σχόλια για το πώς προχωράμε και μετά ο κύριος Φόξ να απαντήσει έτσι και να κάνει μια μικρή περίληψη και να μας επιβεβαιώσει και το χρονοδιάγραμμα βέβαια. Um, Καλημέρα σας. Είμαι ο κύριος Λαντέρο από την ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Παρακολουθούμε τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Ε, αποτιμούμε την ε, έκθεση του κυρίου Μποβέ και διαβάσαμε με ενδιαφέρον το σχέδιο γνωμοδότησης. Θεωρούμε ότι η βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής η βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής ε, συμβανδίζει με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Οκτωβρίου 2009, αλλά στην έκθεση Μποβέ έχουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την ΚΑΠ για το μέλλον. Εξετάζουμε το σχέδιο ε, γνωμοδότησης, το σχέδιο συστάσεων, για να δούμε τι είναι εφικτό και τι όχι, πριν από την ε, τελική μας έκθεση. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μία θέση της Προεδρίας που καλύπτει τα ίδια με το σχέδιο γνωμοδότησης και εστιάζουμε την προσοχή μας στα στις συμβάσεις σε θελούσιας βάσης με βάση τους κανόνες ανταγωνισμού και την οργάνωση της ενίας αγοράς. Αυτά παραμένουν όμως το περιθώριο της ανακοίνωσης του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαντέρο. Κύριε Φόξ, θέλετε να συνοψίσετε. Έχω το χρονοδιάγραμμα ή μπορείτε να το αναφέρετε εσείς. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια. Αυτή είναι η πρώτη ε, γνωμοδότηση για την οποία είμαι υπεύθυνη και με μεγάλη μου χαρά συνεργάστηκα με συναδέλφους ανά την Ευρώπη. Ε, ο κύριος Σμιτ ε, μετά τις 6 Μαΐου θα συνεργαστεί με πιο συντηρητικούς συναδέλφους. Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο γιατί νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα θέματα. Απλώς ανακοινώστε το χρονοδιάγραμμα εσείς. Ευχαριστώ. Απλώς να επιβεβαιώσω ότι έχουμε και ένα σημείωμα για την ε, δημόσια ακρόαση. Κύριε Φόξ, ελπίζω να μπορέσετε να μεταβείτε. Η προθεσμία είναι η 6η Μαΐου για τροπολογίες. 2 ε, Ιουνίου θα τις εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε στις 3 Ιουνίου και στην Επιτροπή Γεωργίας στις 8 ε, Ιουνίου. Θα ήθελα, με βάση τα σχόλια του κυρίου Σμιτ για το κέρδος στον τομέα της Λιανικής, περιμένουμε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για την εποπτεία του τομέα της Λιανικής στις 18 Μαΐου που μπαίνει και στο δικό μας χρονοδιάγραμμα. Στόχος είναι να αναγνωρίσουμε τις λειτουργίες του τομέα της λιανικής από πλευράς προμηθευτών και καταναλωτών. Θα μας απασχολήσει λοιπόν και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί όλα αυτά δεν θα ισχύουν μόνο στον τομέα των τροφίμων της γεωργίας θα υπάρξει αλληλοκάλυψη εργασιών και από την Επιτροπή Άγκρη. Θα ήθελα λοιπόν να μας βοηθήσετε σε αυτή τη συγκρότηση. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Φόξ θα μπορέσει να ασχοληθεί και με αυτά, αλλά θα του αποστείλουμε ένα αντίτυπο και στους σκιώδεις. Ωραία. Θα ήθελα να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο που θα έχουμε μία παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς για το ΣΜΑΣ και αφορά και την έκθεση του Λουί Γκρέχ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Έμερ Ντέιλι που είναι διευθυντής. Έχουμε τις διαφάνειές σας έτοιμες και μπορείτε να αρχίσετε με την παρουσίασή σας. Are you waiting for the system to fire up? Anyway, your slides are here on the computer. We hope that through the magic of technology we may get them up on the screen. Έχουμε τις διαφάνειες έτοιμες. Πρόγραμμα δράσης. Introductory remarks, Mrs. Daly, and then we'll uh, we'll endeavour to get them up on the screen. Uh, so that you can then talk. Ας προετοιμαστούμε και σας δίνω το λόγο για να έχουμε τη δυνατότητα να υποβληθούν και ερωτήσεις. Perfect timing. The miracle of modern technology. Uh, Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much to everybody. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ, γιατί αυτό το πρόγραμμα δράσης είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια, ένα κοινό πρόγραμμα. Πολλοί είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς Μετά από την ε, προηγούμενη αναθεώρηση του 2007 της ενιαίας αγοράς, ε, το Εύρωμα Βαρόμετρο διενέργησε μία έρευνα και είδε ούτε, ότι ούτε οι πολίτες ούτε οι επιχειρήσεις ήξεραν πού να κινηθούν για να λάβουν ε, πληροφορίες για την ενιαία αγορά. Βλέπετε όμως ποιοι είναι οι ιστότοποι και οι άλλες πηγές. Και πέρα από αυτό το συνεφάκι άγνοιας, μεταξύ όλων των, ε, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών δεν ήξεραν τίποτα ε, για διάδραση μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών. Άρα αυτό που κάναμε ήταν να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα ερωτήματα τα διαχειριζόμαστε καλώς. Αυτές είναι πληροφορίες για σας, γιατί πόσο, έχουμε, πόσο μακριά έχουμε κινηθεί. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ο κάθε τομέας ήταν ε, ξεχωριστός και υπήρχε θέμα εδαφικότητας και εδαφικής κυριαρχίας, αν θέλετε. Ένα από τα θέματα που με απασχολεί και εσάς είμαι ευγνώμων είναι ότι μας υποστηρίξατε από πλευράς προϋπολογισμού. Και έτσι μπορέσαμε να συνεργαστούμε με αυτές τις υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα δράση υπάρχουν τρία, τρεις διαφορετικοί τομείς. Καταρχήν η καλύτερη πληροφόρηση, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καλύτερα, έτσι ώστε αυτό να γίνει αποδεκτό από τους πάντες, καλύτερη θέση σε ισχύ, έτσι ώστε να υπάρχει καλή λειτουργία και ενδεχόμενη επίλυση προβλημάτων. Και το πιο ενδιαφέρον για μας και για σας είναι να έχουμε ε, αποδείξεις από αυτή την, κυψέλη δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αναλάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες οι οποίες να βασίζονται σε αποδεκτικά στοιχεία που λαμβάνουμε. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες. Καλύτερες ε, πληροφορίες έτσι ώστε να μπούμε σε ένα νέο τομέα ιδιόγλωσσας κατά κάποιο τρόπο και να υπάρχει ένα ε, ενίο σημείο εισδοχής το οποίο να είναι διαχρονικά διαθέσιμο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. Βασίζεται σε οκτώ διαφορετικούς τομείς που είναι οι τομείς που κατά τη γνώμη μας ε, λειτουργούν με βάση τις ε, πληροφορίες που λαμβάνουμε για την εσωτερική αγορά. Τομείς που έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις, γιατί είναι θέματα που τις απασχολούν. Εδώ είναι ε, μια θεματική που βασίζεται στην προσέγγιση του χρήστη. με βάση την κινητικότητα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα από τη ζωή. Δηλαδή μικρές ιστορίες ε, με καλό τέλος και όχι κακό. Έτσι ώστε να δείξουμε στους πολίτες τι μπορεί πραγματικά να συμβεί. Επίσης υπάρχει διάδραση έτσι ώστε να έχουμε feedback, να έχουμε ανάδραση. Έτσι ώστε όταν έχουν προβλήματα οι πολίτες να καλύπτονται, να μας δίνουν δηλαδή να υπάρχει διαδικασία ανάδρασης. ακούμε τους πολίτες και μπορούμε να τους παραπέμψουμε και σε άλλες υπηρεσίες εκεί που μπορούμε. Πού βρισκόμαστε τώρα. Βρισκόμαστε μεσοστρατής. Η ανάδραση είναι πολύ ενθαρρυντική, υπάρχει στα αγγλικά, αλλά θα δούμε αυτή την ε, ε, διάδραση σε ε, όλες τις γλώσσες για να υπάρξει μια εκστρατεία για όλους. Προκλήσεις. Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις. Για να είναι επικαιροποιημένη η πληροφόρηση θα πρέπει να βασιστούμε στα κράτη-μέλη διότι πρέπει να κατέβουμε στο πεδίο των κρατών μελών και αυτή είναι η πρόκληση που θα πρέπει να μας απασχολήσει και νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Εργαζόμαστε με τις εθνικές διοικήσεις και κυβερνήσεις. Γιατί αν δεν είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία, δεν είναι χρήσιμα. Αν ξέρουμε πως έχει κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη, βλέπουμε κατά πόσο υπάρχουν ε, λανθασμένες ροές στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Το γλωσσικό είναι αδύσβατο θέμα. Θα πρέπει να καλύψουμε όλες ε, τις γλώσσες έτσι ώστε να έχουμε ποιοτική εργασία. καλύτερη εφαρμογή. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη προσπελασιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες αρρωγής. Υπάρχει το πεδίο Solvit μετά από τις συζητήσεις σας. Και τώρα εργαζόμαστε με τις ε, διάφορες υπηρεσίες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν ε, ιστό, έναν δίκτυο διάδρασης και να βρούμε νέους τρόπους συνεργασίας. έτσι ώστε να δίνουμε συμβουλές πρόσωπο με πρόσωπο και να έχουμε, να προβάλλουμε και εργασίες ε, ενσυνειδητότητας. Το Solvit ε, απαρτίζεται από προσωπικό από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μεγάλη λιτότητα ως προς τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα πρόβλημα και χώρου και χρόνου και χρήματος δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη εργασία για τα κέντρα Solvit και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της ε, νομικής, των νομικών συμβουλών και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προβάλλουμε συνέργειες ο το δίκτυο των εθνικών διαμεσολαβητών θα μπορούσε να ήταν το σωστό δίκτυο προβολής συνεργειών. Τώρα, καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό μας ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Διενεργούμε μία πιλωτική έρευνα φέτος Παίρνουμε αποδεικτικά στοιχεία από πέντε κέντρα αρρωγής να δούμε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε από αυτά τα μικροτομεακά προβλήματα. Θα δούμε είναι το, ποια είναι τα αποτελέσματα και θα τα αναλύουμε και ως προς τα επαγγελματικά προσόντα είναι κάτι το οποίο θα παρουσιάσουμε στο, επόμενο scoreboard. Στο επόμενο βαθμολόγιο. Άρα τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι κρίκοι που λείπουν θα πρέπει να καλύψουμε όλους τους τομείς και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα μαζί σας. Νομίζω λοιπόν σας δώσαμε μία πρόγευση της κατάστασης και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όλη σας την υποστήριξη, τη μέχρι τώρα υποστήριξη και ίσως αυτό να δημιουργήσει μεγαλύτερη εργασία και συνέργειες μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Ο Λουί Κρέγκ κάθεται δίπλα μου και υπάρχει η έκθεση κυρίας Twins που σχετίζεται με την εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να συνδράμουμε με βάση τη Single Market Act, την πράξη ενίας αγοράς. Και ο Λουί Γκρέκ και εγώ το συζητάμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό βήμα προς τα μπρος. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο. Um, um, Ποιοι θέλουν το λόγο. So I'll give Mrs. the floor first. Έχετε το Um, thank you very much. Um, at last, this initiative. I mean... Επιτέλους, ήρθε η ανακοίνωση. Εγώ δούλευα κάποτε στην ε, Κομισιόν και ήμουν εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Πολωνία και από τότε Ονειρευόμουν να υπάρξει έτσι μια διεύθυνση που να μπορεί κανείς να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Και θυμάμαι ότι κάθε πρωτοβουλία, το Solvit, το Euronews κτλ. ξεκινούσε από τις αντιπροσωπείες, πλήρως λειτουργική, με τα ε, με τις πληροφορίες και εγώ δεν μπορούσα, δεν είχα χώρο στην ιστοσελίδα μου να βάλω όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και επιτέλους έχουμε τώρα μια τέτοια σελίδα η οποία επιτρέπει σε μια διεύθυνση να βρίσκει κανείς ό,τι θέλει, να ανοίγει τις σελίδες, να πηγαίνει στο βάθος των πραγμάτων. Ελπίζω με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο να συνεχίσετε. Να είναι καλή η συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες σας στην Κομισιόν και αυτό είναι πρόκληση καμιά φορά. Εμείς θα κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη μας για να σας δώσουν το feedback που χρειάζεστε και τις πληροφορίες και θα το προωθήσουμε όλοι μαζί. Αναφέρατε το φόρουμ για την ενιαία αγορά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια πολύ καλή πλατφόρμα για να προωθήσουμε για να ενημερώσουμε τους πολίτες για όλες αυτές τις πηγές πληροφόρησης, ώστε όχι απλώς να βλέπουν τι είναι ωφέλιμο για αυτούς από την Ευρώπη και από την ενιαία αγορά, αλλά θα μπορούν να το χρησιμοποιούν κιόλα. Και αυτό θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στη λειτουργία της εσωτερική ενιαίας Και εκεί εμπλέκονται και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Κάναμε την ε, μεγάλη συζήτηση σήμερα για την Ευρώπη των πολιτών και, των, ε, και τις επιχειρήσεις. Οπότε εδώ στο φόρουμ δείχνουμε ότι γίνεται να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Ε, για την ξύλινη γλώσσα που είπατε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, και εγώ συμφωνώ. Ειδικά με, τις, με τα κρονίμια που κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα ποτέ και δεν ξέρει και από ποια γλώσσα προέρχονται. Επίσης, το φθινόπωρο θα γίνει ένα φόρουμ για την ε, νέα αγορά, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να ενισχυθούμε και οι δύο από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για τη δουλειά που κάνατε και για τη συμβολή σας. Άλλος κανείς. Εγώ σύντομα να κάνω ένα σχόλιο και να θέσω ένα ερώτημα. Το να υπάρχει αυτή η κοινή πύλη είναι όντως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι η διαφορά σε ό,τι αφορά το branding και την ε, θέση σε εμπορία και τους πολίτες μου φαίνονται σαν να μπλέκουν λίγο τους πολίτες. Το Your Europe είναι το εργαλείο που σας δίνει το Europe Citizens για να προχωρήσετε θέλετε να κάνετε κάποιες στοχοθετημένες εκστρατείε, αλλά πριν προωθήσετε οτιδήποτε, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβετε κάποιες ε, συμβουλές ό,τι αφορά τη θέση σε εμπορία, πώς δηλαδή μπορείτε να το πουλήσετε το αντικείμενο και το προϊόν σας αυτό. Και δεύτερον, για το Euro for Citizens, δεν είναι απόλυτα σαφές πού θα αποταθώ εγώ αν έχω προβλήματα ως καταναλωτής αν έχω πρόβλημα με μια υπηρεσία ή με ένα προϊόν, πού πάω. Ίσως να υπάρχει ξεχωριστό, ξεχωριστή σελίδα γι' αυτό. Αλλά με βάση και, με το, και το ότι επικεντρωνόμαστε στον, ε, στους ε, καταναλωτές και έχουμε πρόσβαση στα προβλήματα των καταναλωτών, και στις υπηρεσίες που ε, προσφέρουν ε, οι ε, ενώσεις καταναλωτών και που μιλούμε και για ποιότητα υπηρεσιών και για διασυνοριακές υπηρεσίες, είναι θέμα ποιότητας τελικά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών μπορούν να συνδεθούν με αυτό το πόρταλ, με αυτή την πύλη. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα διαφορετικό εμπορικό όνομα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες πολύ καλές ιδέες και προωθούν την όλη ιστορία. Αλλά το SMAS, όπως είπε και η κυρία Τούνσεντ, ε, είναι άλλο ένα ακρονίμιο. Ε, τώρα το SMAS ε, δεν είναι και πολύ έβυχο. Οπότε μην το χρησιμοποιήσετε αυτό στο μέλλον. Σκεφτείτε κάτι πιο δυναμικό ίσως και πιο φιλικό προς το χρήστη. I've now finished my contribution from my, but I, so I know as chairman. Οπότε έχετε το λόγο τώρα για να, απο, να απαντήσετε και στην κυρία Τόνσεν και σε εμένα. Uh, well, thank you very much. Σας ευχαριστώ. To Mrs. Van Thun. I... Ευχαριστώ κυρία work... Είναι πρόκληση για μας να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αν δείτε την ομοθέσια περί ενιαίας αγοράς και όλες τις διαφορετικές πτυχές, έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς, 14 διαφορετικούς φόρεις. Επειδή όμως έχουμε αγαστές σχέσεις, ε, εντάξει, δεν πειράζει. Βεβαίως, αν χρησιμοποιήσουμε το φόρουμ ε, προαγωγής, αυτό είναι ένα, μια, μια κατάσταση ολικού κέρδους. Ένα από τα στοιχεία που θα ήθελα να αναφέρω σε σχέση με την ε, αποφασιστικότητά μας θα θέλαμε να ασχοληθούμε και με τις επιχειρήσεις γιατί από πλευράς επιχειρήσεων υπάρχει μια αποδόμηση ως προς το ενδιαφέρον και για ε, μια πύλη εσωτερικής αγοράς αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα ιδίωνο θα πρέπει να προωθήσουμε και την ε, πλευρά των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση για μας. Γιατί μιλήσαμε με εμπορικά επιμελητήρια, με διάφορα πάνελ, με όλο, όλο το, το, το πλαίσιο, τον επιχειρηματικό κόσμο και σε σχέση με τα σήματα και την απλούστευση, αυτή είναι και η απότερη πρόκληση. Διότι σας δείξαμε το περιεχόμενο, αλλά εάν θέλουμε να μπούμε στη συνολική λογική, θα πρέπει να απλουστεύσουμε σε σχέση τώρα με τα προϊόντα που θέλουμε Θέλουμε να έχουμε έναν αριθμό, μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτά τα στοιχεία θα αποσταλούν στο σωστό σημείο. Ο καθένας θέλει το δικό του σήμα. Τώρα το SMAS δεν είναι σήμα, δεν είναι brand name, είναι ένα ακρόνιμο μεταξύ μας για το τι κάνουμε. Γι' αυτό θα ενταχθεί στο, ε, μάλλον θα, θα ενταχθεί στη δική μας λογική, αλλά θα φύγει από την γενικότερη ορολογία. Γιατί θέλουμε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτό αποτελεί πρόκληση. Προσπαθούμε λοιπόν να μπούμε δυναμικά σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος για την προσέγγιση σας, για την ανοιχτή σας προσέγγιση. Θα λάβετε υπόψη τα σχόλιά μας. Είναι επικοδομητική κριτική γιατί δεχόμαστε ε, την εργασία σας είναι ευπρόσδεκτη στα πλαίσια του Single Market Act έτσι ώστε να προβάλλουμε προτάσεις φιλικές προς το χρήστη. Και έτσι τα κράτη-μέλη μπορούν να υποστηρίξουν και το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Υπάρχει πολύ καλή εταιρική σχέση. Σας ευχαριστώ. Σας υπενθυμίσω ότι το απόγευμα θα συναντηθούμε στην 4Q1 στις 3 ε, για την διακοινοβουλευτική συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την εσωτερική αγορά ως προς ε, τις υπηρεσίες. Ελπίζω να μπορέσατε να συνεισφέρετε όλοι και θα ξαναβρεθούμε εδώ αύριο το πρωί. Άρα τα στοιχεία, τα έγγραφά θα μεταφερθούν. Ο κύριος Μπαρνιέ θα είναι εδώ στις 9 και στις 10 και 4 θα ψηφίσουμε. Μην ξεχάσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα χέρι.